να διεκπαιρεώσουμε το σημείο που αφορά την έγκριση με διάταξη αν δεν έχετε αντιρρήσει και να σας ενημερώσω εν συντομία δυνάμει των κανόνων που έχουμε σε σχέση με τους ε, τριμερείς διαλόγους που είναι σε εξέλιξη. Όπως γνωρίζετε εργαζόμαστε πολύ σκληρά για το τραπεζικό πακέτο προκειμένου να έχουμε ολοκληρώσει. Όχι μόνο να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και να έχουμε στο δυνατόν νωρίτερα κάποια συμπεράσματα για να συμβάλλουμε τα μάλα στις σημαντικές συζητήσεις ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πριν ε, αυτού βέβαια του ΕΚΟΦΗΝ για τη μεταρρύθμιση της ΩΝΕ και τα διάφορα στοιχεία του πακέτου. Θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές, τους κοιόδης, καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για να οριστικοποιηθούν τα βασικά στοιχεία αυτού του πακέτου. Στις 22 Νοεμβρίου είχαμε τον 7ο τριμερή διάλογο για τον κανονισμό και την οδηγία για τις κεφαλακές απαιτήσει, το CRRD και το CRRD5. Καταφέραμε να σημειώσουμε συμφωνία σε θέματα που αφορούν την αναλογικότητα, το δίκτυο καθαρή σταθερή χρηματοδότηση, ε, το πιστοτικό κίνδυνο, trading book, η διακεφάλαια, intermediate parent undertaking, το ποσοστό μόχλευση ε, και θα χρειαστεί να ολοκληρώσουμε κάποια άλλα σημεία. Δεν έχουμε ακόμη οριστικό κείμενο για όλα. Θα προσπαθήσουμε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Είχαμε επίσης ε, στις 21 Νοεμβρίου <clears throat> και μέσα στη νύχτα ε, τον έκτο τριμεριδιάλο για τον BRD με τον ίδιο στόχο. Να ολοκληρώσουμε τα πιο σημαντικά. Και κοντεύουμε. Έχουμε καταλήξει σε προσωρινή συμφωνία που θα εξαρτηθεί από την επίλυση κάποιων άλλων ζητημάτων σε ό,τι αφορά το subordinated debt. για το moratorium, για τις υποχρεώσεις, bail, liabilities κτλ. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν τα κρατημέλη και πώς θα ολοκληρωθούν και οι άλλες πτυχές για να δούμε το συνολικό πακέτο. Είχαμε και τον πρώτο τιμερή διάλογο για τις διασυνορικές πληρωμές ΣΕΠΑ, 19 Νοεμβρίου. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως ξέρετε, δεν συμφωνούσαν σε αυτό το παιδί πρότασης. Εμείς θέλουμε τα ίδια τέλη χρέωσης να ισχύουν για, όλες τις, για τα νομίσματα, ενώ μόνο σε μεταφορές σε ευρώ θέλει να ισχύει αυτό το Συμβούλιο, όπως και η Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, επί της αρχής το Συμβούλιο συμφωνεί με τη θέση του Κοινοβουλίου. Απλά δεν ξέρουμε ακριβώ τι γίνεται με τους ε, παρόχου υπηρεσιών που μάλλον ε, θα επιμεριστούν ανάλογο βάρο. Υπάρχουν και κάποια άλλα μη πολιτικά θέματα. Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ε, ο επόμενος τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για την εβδομάδα της 3 η Δεκεμβρίου. Και μετά από όλα αυτά μπορούμε να περάσουμε στον δημοσιοματικό διάλογο με τον κύριο Ντράγκη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στη συνέχεια θα μας μιλήσει υπό διαφορετική ιδιότητα. Πρώτα όμως ως πρόεδρος της ΕΚΤ και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντράγκη που είστε εδώ. Πολύ κρίσιμη, σημαντική χρονική στιγμή πριν την αποφασιστική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δεκεμβρίου. σημειώνουμε και επικροτούμε την πρόσφατη απόφαση που έλαβε η ΕΚΤΑ Ίσως έχουμε ανάλογα με τα δεδομένα βέβαια μια σημαντική απόφαση το Δεκέμβριο, αλλά αν ε, κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα ε, τις δηλώσεις στο κείμενο που έχετε συντάξει, φαίνεται ότι έχετε δεσμευθεί να ακολουθήσετε μια νομισματική πολιτική και μετά τον ε, Δεκέμβριο που θα είναι αρκετά υποβοηθητική και αυτό είναι σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη τη μακροοικονομική κατάσταση και τις προκλήσεις που θα συζητηθούν φαντάζομαι και στη διάρκεια της ακρόασης. Έχουμε αυτή την ε, τελμάτωση με την έλλειψη ανάπτυξης, χαμηλά επιτόκια, ονομαστικά και πραγματικά. Τέλος πάντων έχουμε διάφορα θέματα που μας απασχολούν και έχουμε σχετικά έγγραφα, καταθέσει. Ξέρουμε ότι έχει κάνει στη εξτηρευστότητα για την επίτευξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών και υποφασιστικός ρόλος της ΕΚΤ είναι γνωστός επίσης και για την υποστήριξη του ευρώ. Θα σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που είστε εδώ και θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές ε, της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι στην Επιτροπή σας για την τελευταία ανταλλαγή απόψεων του έτους. Έχετε επιλέξει πολύ επικαιρά ζητήματα για τη σημερινή μας συζήτηση. Οπότε θα ξεκινήσω αμέσως και θα μπω στην ουσία. Πρώτα απ' όλα, θα σας πω ποια είναι η αξιολόγησή μας για την οικονομική προοπτική της Ευρωζώνης και το τι σημαίνει αυτό για την νομισματική μας πολιτική. Δεύτερον, θα συζητήσω γιατί ο σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στην ΟΝΕ θα στηρίξουν την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και άρα την οικονομία της Ευρωζώνης. Τα δεδομένα τα οποία ε, προέκυψαν από την τελευταία μου επίσκεψη εδώ τον Σεπτέμβριο ήταν κάπως ασθενέστερα από ό,τι περιμέναμε. Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,2% στο τρίτο τρίμηνο αυτό ακολουθεί την αύξηση του 0,4% στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2018. Η ανάπτυξη επιβραδύνεται και αυτό οφείλεται κυρίως στην χαμηλότερη ανάπτυξη του εμπορίου αλλά και σε κάποιους παράγοντες που οφείλονται σε συγκεκριμένες χώρες και κλάδους. Θεωρούμε τώρα ότι αυτή η επιβράδυνση είναι προσωρινή ή πιο μακροπρόθεσμη. Μια σταδιακή επιβράδυνση είναι φυσιολογική καθώς ε, η επέκταση, η πιστοτική και η ανάπτυξη συγκλίνουν. Μάλιστα, ως ε, προς το μέλλον αναμένεται να μειωθεί η αύξηση της ανάπτυξης ε, καθώς θα έχουμε κάποιες μικρότερες ελλείψεις στην προμήθεια εργασίας. Επίσης θα ομαλοποιηθούν και τα ποσοστά αποταμιεύσεων. Αυτά φαίνονται και στις ε, προβλέψεις μας ε, του Σεπτεμβρίου που προβλέπουν ετήσια ανάπτυξη 2,0% και μετά ελαφρώς ε, χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξη 1,8% το 19 και 1,7% το 2020. Κάποια από αυτή την επιβράνηση ίσως είναι προσωρινή. Μάλιστα τα πιο τελευταία δεδομένα δείχνουν μια ομαλοποίηση της παραγωγής στην αυτοκίνητο βιομηχανία που είχε αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω παραγόντων οι οποίοι ήταν παράγοντες οι οποίοι εμφανίστηκαν άπαξ. Επιπλέον, καθώς σταθεροποιείται και το παγκόσμιο εμπόριο, θα μπορούσε επίσης και αυτό να έχει μόνο προσωρινές επιπτώσεις. Ταυτόχρονα υπάρχουν όμως κίνδυνοι σε σχέση με τον προστατευτισμό, τις ευπάθειες της αναδυόμενες αγορές και την κινητικότητα στις χρηματαγορές και βεβαίω ε, τα βασικά της εγχώριας ζήτησης παραμένουν σταθερά. Το εισόδημα των νοικοκυριών συνεχίζει να υποστηρίζεται από υψηλά επίπεδα χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων και περαιτέρω βελτιώσει στην αγορά εργασία. Το ποσοστό ανεργία μειώθηκε στο 8,1% τον Σεπτέμβριο του 2018, το χαμηλότερο επίπεδο δηλαδή που έχει παρατηρηθεί από το τέλος του 2008 και η απασχόληση συνεχίζει να αυξάνεται στο τρίτο τρίμηνο επιπλέον. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων υποστηρίζονται από τις πολύ ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες στην Ευρωζώνη μαζί με την σταθερή ζήτηση και την αυξανόμενη κερδοφορία. Όσον αφορά τις εξελίξεις των ε, τιμών, ο συνολικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,2% τον Οκτώβριο φέτος από 2,1% τον Σεπτέμβριο τα μέτρα του βασικού πληθωρισμού εξακολουθούν να είναι χαμηλά αλλά έχουν αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Γενικά υπάρχει λόγος να πιστεύουμε πως ο βασικός πληθωρισμός θα αυξηθεί σταδιακά την περίοδο που έρχεται. Οι μισθοί αυξάνονται καθώς ε, συνεχίζουν να βελτιώνονται οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και οι λήψεις ε, σε κάποιες ε, χώρες. Αναμένεται επίσης ε, αύξηση των μισθών, η οποία θα συνεχίσει να στηρίζει την προσαρμογή προς τα άνω του βασικού πληθωρισμού. Επιπλέον, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες των αγορών και του πληθωρισμού είναι γενικά καλά εδρεωμένες και συμφωνούν με αυτήν την προοπτική. Συνολικά, οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προηγούμενες αξιολογήσεις του ΔΣ της Τράπεζας για τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό και συνεχίζουν να στηρίζουν την πεποίθησή μας ότι η σύγκληση του πληθωρισμού με των στόχων μας θα συνεχιστεί και θα διατηρηθεί ακόμα και μετά την σταδιακή μείωση των αγορών στοιχείων ενεργητικών από την τράπεζα. Οπότε το ΔΣ συνεχίζει να θεωρεί ότι υπό την αίρεση της επιβεβαίωση της, προβλε... της μεσοπρόθεσμης πρόβλεψής μας από τα δεδομένα, οι αγορές αυτές θα τερματιστούν τον Δεκέμβριο του 2018. Ταυτόχρονα οι αβεβαιότητες εξακολουθούν να απαιτούν υπομονή και συνέπεια και συνέπεια στον υπολογισμό της νομισματικής μας πολιτικής. Απαιτείται ακόμα ένα νομισματικό κίνητρο για να στηρίξουμε την περαιτέρω αύξηση των ε, εγχώριων πιέσεων τιμών για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να κινείται προς τον στόχο μας ε, θα διατηρηθεί ένα σημαντικός βαθμός νομισματικού κινήτρου ακόμα και μετά το τέλος του προγράμματος αγορών. Και αυτό θα γίνει βεβαίως ε, και με βάση τις κατευθύνσεις ε, που έχουμε δώσει όσον αφορά την κίνηση των επιτοκίων και από τα αρκετά σημαντικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία έχουμε ήδη αγοράσει και τις ε, σχετικές επανεπενδύσεις. Τώρα να αφαιρθώ στην μεταρρύθμιση της ΟΝΕ. Για να μείνω στα θέματα τα οποία έχετε επιλέξει για τη σημερινή συζήτηση, να εξηγήσω γιατί μια πληρέστερη ΩΝΕ θα στηρίξει την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, θα αναφερθώ σε δύο είδη προκλήσεων που προκύπτουν σε μια ΟΝΕ η οποία δεν είναι ολοκληρωμένη όπου η νομισματική πολιτική είναι όντως ευρωπαϊκή ενώ άλλα σημαντικά τμήματα της οικονομικής πολιτικής παραμένουν στο εθνικό επίπεδο πρώτον η Ευρωζώνη είναι εκτεθειμένη σε κραδασμούς που προκύπτουν από παγκόσμιους κραδασμούς ή κοινέ ευπάθειες. η κοινε ευπαθειες οικονομική κρίση του 2007 και 2008 και τα επακολουθά τους ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα καθώς η ανάπτυξη πέρασε σε αρνητικό ρυθμό σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης το 2009. Αυτό το οποίο έκανε την Ευρωζώνη διαφορετική από τις άλλες οικονομίες ήταν το ότι δεν υπήρχε μια δημοσιονομική ικανότητα για ολόκληρη την Ευρωζώνη για να συμπληρώσει την νομισματική πολιτική. Επιπλέον, δεν υπήρχε ένα εύρωστο ρυθμιστικό εποπτικό πλαίσιο διαχείρισης των κρίσεων όταν ήρθε η κρίση και έτσι αυξήθηκαν οι αμφιβολίες για την ευρωστία του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Αυτό με τη σειρά του επηρέασε την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και την μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Δεύτερον, όπως είδαμε και στην προηγούμενη κρίση, η Ευρωζώνη είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που προκύπτουν από εγχώριες πολιτικές οι οποίες καταλήγουν σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα χρέους, σε ευπάθειες του χρηματοπιστωτικού τομέα και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Μέσω των διάβλων αυτών του χρηματοπιστωτικού, της εμπιστοσύνης και του εμπορίου μπορεί η κίνδυνοι αυτοί να διαχειριστούν σε άλλες χώρες που έχουν στενές ε, διασυνδέσεις ή παρόμοια ευπάθεια με την χώρα από όπου ξεκίνησε ο κίνδυνος. Επίσης, τέτοιες ε, πολιτικές μπορούν να κατακαιρματίσουν τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες, εμποδίζοντας έτσι την ομοιογενή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μας σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και οι πολιτικές αυτές, οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν μακροπρόθεσμα, τελικά καταλήγουν σε κοινωνικά οδυνηρές και χρηματοπιστωτικά ακριβές οικονομικές προσαρμογές που μπορούν να υπονομεύσουν την συνοχή της ΩΝΕ. Εν ολίγης, μία μη ολοκληρωμένη ΩΝΕ έχει αντίκτυπο στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στο οποίο διεξάγουμε την οπισματική πολιτική μας. Η Ευρώπη το μάθημα αυτό το έμαθε με τον σκληρό τρόπο και έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στο να γεφυρώσουμε τα κενά στην αρχιτεκτονική της ΩΝΕ. Παραδείγματος χάρη, Έχουμε τώρα ένα πολύ ισχυρότερο και ολοκληρωμένο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής ρύθμισης, εποπτείας και επίλυσης κρίσεων. Εσείς παίξατε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και το πλαίσιο αυτό επίσης μας βοήθησε να περιορίσουμε οποιονδήποτε κίνδυνο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μπορεί να προκύψει κατά μία περίοδο χαμηλών επιτοκίων. Αλλά πρέπει και μπορεί να σημειωθεί περισσότερη πρόοδο και θα ήθελα να αναφέρω τρει τομεί, όπου απαιτείται να γίνει αυτό. Πρώτον, ένα αποτελεσματικό σύστημα συντονισμού τη πολιτική για να προωθηθούν οι ορθές εθνικέ πολιτικές, μειώνοντα έτσι τι εγχώριε πηγέ τέτοιων κρατασμών και αυξάνοντας την ικανότητα των χωρών να απορροφήσουν τέτοιου κρατασμού όταν αυτοί υλοποιηθούν. Αυτό αφορά την προώθηση χρηστών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών. Γι' αυτό θα πρέπει να αναζωπυρώσουμε την πίστη στους κοινού κανόνες μας και να διασφαλίσουμε ότι γίνονται σεβαστοί. Η επιπλέον στήριξη από το ενωσιακό επίπεδο, όπως πρότεινε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να είναι εποφελής στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων των μεταρρυθμίσεων που τονίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εάν οι οικονομίες Ευρωζώνης είχαν μεγαλύτερα επίπεδα ανθεκτικότητας, θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε έναν κοινό κρατασμό με παρόμοιο τρόπο, μειώνοντας έτσι τις πολύ άκριβες μακροοικονομικές αποκλίσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ενιαία νομισματική πολιτική μας. Η ανάπτυξη τέτοιων υγιών οικονομικών δομών και θεσμών επίσης θα αύξανε την ε, δυνητική παραγωγή. Δεύτερον, όπως πρότεινε πρόσφατα η τράπεζα στη γνωμοδότησή της για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας, η Ευρωζώνη χρειάζεται ένα δημοσιονομικό εργαλείο για να διατηρηθεί η σύγκληση απέναντι σε μεγάλους εξωγενείς κραδασμούς, στηρίζοντας έτσι την ενιαία νομισματική πολιτική μια τέτοια λειτουργία θα πρέπει να εστιάσει στις κυκλικές εξελίξεις και θα πρέπει να είναι υπό την αίρεση ορθών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών σεβόμενοι πλήρως το πλαίσιο διακυβέρνησης της Ένωσης. Αυτό με τη σειρά του θα συνεισέφερε στη μακροοικονομική σταθερότητα στο επίπεδο της Ευρωζώνης και το κυριότερο σε κάθε κράτος μέλος. Και έτσι θα μπορούσε να ληφθεί η δράση πριν χρειαστεί να καταφύγουμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για τις καταστάσεις όπου υπάρχει μια αστάθεια στις αγορές, ο μηχανισμός σταθερότητας παραμένει κέριος για να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της μετάδοσής της. Πρέπει λοιπόν ο μηχανισμός να έχει τα μέσα εκείνα που είναι απαραίτητα για να πετύχει τους στόχους του και να στηρίξει την Τραπεζική Ένωση. Άρα, καλωσορίζω τις συζητήσεις ε, για να γίνει πιο αποτελεσματικός ο μηχανισμός όπως επίσης αναφέρονται σε μια γνωμοδότηση της έκτεπη του θέματος. Τέλος, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η οικοδόμηση μιας ένωσης Κεφαλαιαγορών έχουν ουσιαστική σημασία. Εάν θέλουμε να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, πρέπει να ενισχύσουμε την αντοχή και την ολοκλήρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα βελτιώνοντας έτσι και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μας. Βεβαίω. αυτά τα οποία είπα θα στήριζαν την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, όμως δεν είναι αυτό το μόνο όφελος. Το κυριότερο κίνητρο για αυτές τις πρωτοβουλίες θα είναι να δουν απτά ωφέλη από το κοινό νόμισμα όλοι οι Ευρωπαίοι. Η στήριξή τους για το ευρώ έχει αυξαθεί καθώς η ΟΝΕ ανακάμπτει από την κρίση και τώρα βρίσκεται σε ένα ιστορικό υψηλό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα απογοητευτούν. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες, μέχρι το τέλος αυτής της θητείας, οι ημέρες αυτές θα είναι αποφασιστικές για να σημειωθούν συγκεκριμένα βήματα στη μεταρρύθμιση της ΟΝΕ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως παίξει έναν κρίσιμο και επικοδομητικό ρόλο έτσι ώστε οι συζητήσεις αυτές να εστιάσουν σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση και στην οικοδόμηση αποτελεσματικών κοινών θεσμικών οργάνων. Ξέρουμε πως η μετάβαση από τον συντονισμό στην κοινή λήψη αποφάσεων από κοινού κανόνες σε θεσμικά όργανα είναι αναγκαία, αλλά απαιτεί χρόνο. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για αδράνεια πολλά από τα βασικά βήματα πρέπει να γίνουν τώρα. Δηλαδή να σχεδιαστεί ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των μερών. Είμαι πεπισμένος πως εσείς και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παίξετε και πάλι ένα κέριο ρόλο στην προώθηση αυτού του προγράμματος της ΟΝΕ έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα στην 20η επέτειο του ευρώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι τώρα στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Thank you Ευχαριστούμε πολύ. President Draghi. Πολύ συμμεριζόμαστε αυτό που είπατε στο τέλος ε, της παρέμβασή σα, ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνη ε, και ο σχεδιασμός ενός φιλόδοξου σχεδίου μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμη σημασία. Πρόσφατα το Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι το 74% των Ευρωπαίων στηρίζουν, μάλλον των κατοίκων της Ευρωζώνης, στηρίζουν το ευρώ που είναι ρεκόρ από το 2002 και νομίζω ότι αυτή είναι και μεγάλη συμβολή ε, και αξία του έργου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τη στήριξη της αξιοπιστίας της Αν θέλουμε όμως ε, να συνεχιστεί αυτή η τάση και να είμαστε και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τυχόν μελλοντικέ κρίσει, πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο και σε ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει. Γι' αυτό είναι σημαντική και η δική σα έκκληση και εμεί είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε αυτό το εγχείρημα. Αναφερθήκατε προηγουμένω ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίηση Επενδύσεων, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για μένα. Α περάσουμε τώρα στι παρεμβάσει των μελών. Ο κύριος Κίρτσος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράγκη, συμφωνώ με την ανάλυση σας. Όμως μου φαίνεται ότι υπάρχουν προκλήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει μία Ω ως προς τις μεταρρυθμίσεις σε ορισμένες ε, χώρες της και έχουμε και δύσκολες ευρωεκλογέ μπροστά μας. Πιστεύετε ότι μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που περιγράψατε παρά το γεγονός ότι όσο πολιτική ε, αναγκαστικά ε, θα πρέπει να εξετάσουμε και την πολιτική σκοπιά εν ώψη και των ευρωεκλογών. Πώς γίνεται λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή την τροχιά που περιγράψατε, γιατί εμείς ως πολιτικοί πρέπει να κάνουμε και πολιτικούς υπολογισμούς εν ώψη των ευρωεκλογών. Για παράδειγμα, έχετε την κατάσταση στην Ιταλία. Διάβασα την κριτική της ε, Κεντρική Τράπεζα ε, τη Ιταλία προ την Ιταλική κυβέρνηση, αλλά τελικά ποιο θα αποφασίσει τι θα γίνει. Και ένα δεύτερο ερώτημα για τον Brexit γνωρίζουμε τους όρους της συμφωνίας. Πιστεύετε ότι συνδέεται ένα κόστος εδώ σε ό,τι αφορά την ε, δομή, τη χρηματοοικονομική δομή της Ευρωζώνης και αν το Βρετανικό Κοινοβούλιο απορρίψει τη συμφωνία. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β. Τι θα γίνει τελικά στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ και τα δύο ερωτήματα που θέσατε είναι αρκετά δύσκολα. Με ρωτήσατε αρχικά αν η κατεύθυνση στην οποία εγώ σας λέω ότι πρέπει να κινηθείτε ε, είναι εφικτή δεδομένης της συγχρονική συγκυρίας. Είναι εφικτή, είναι ρεαλιστική. Ε, απαιτεί φυσικά ένα φιλόδοξο όραμα και αποφασιστικό ε, αυτοπεποίθηση και πίστη στο κοινό μας όραμα. Και πιστεύω ότι αυτό το όραμα γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή ευρύτερα είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι συμμερίζονται. Τώρα υπάρχουν ε, ε, ειδικέ καταστάσεις ανάλογα και με τη χώρα και με τις περιστάσεις που τα πράγματα φαίνονται πιο δύσκολα αλλού λιγότερο. Θα δούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα ένα εφικτός στόχο, μια εφικτή κατεύθυνση. Και πάλι και το δεύτερο ερώτημά σα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Τι θα γίνει σε περίπτωση αρνητικού σεναρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα, η ΕΚΤ, η Αγγλική ε, Κεντρική Τράπεζα και η Βρετανική Κυβέρνηση τα έχουν συζητήσει και μάλιστα η ΕΚΤ και η Βρετανική Κεντρική Τράπεζα εργάζονται από κοινού. Ε, εντοπίζουμε λοιπόν ε, τα βασικά προβλήματα, τις βασικές ευπάθειες που μπορούν να προκύψουν από απότομη ε, επιδείνωση των πραγμάτων. Μπορώ να σας πω ότι γενικά, ιδίως μετά την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε προσφάτως, οι περισσότερες ε, από αυτές τις αβεβαιότητες ε, μπορούν να αντιμετωπιστούν ε, επαρκώς και να μην διακινδυνευτεί έτσι η σταθερότητα. Η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στην πρόταση της Κομισιόν ώστε τελικά να δημιουργηθεί εμβριακά στο μια λειτουργία σταθεροποίησης ε, στην Ευρωζώνη και έχετε γνωμοδοτήσει θετικά τη βλέπουμε στη γνωμοδοτησή σας αν και κάποιες πτυχές της ε, πρότασης της Κομισιόν ε, σας βρίσκουν αρκετά επιφυλακτικούς. Επιμείνατε όμως και στη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτής της σταθεροποιητικής ε, λειτουργίας και των δημοσιονομικών κανόνων και του Συμφώνου Σταθερότητας. Μήπως υπάρχει αντίφαση. Απ' τη μία δηλαδή να υπάρχει αυτή η σταθεροποιητική λειτουργία και από την άλλη να απαιτείται πλήρης σεβασμός στους δημοσιονομικούς κανόνες. Και καταλαβαίνετε γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε μια χώρα η οποία πλήττεται από ασύμετρους κραδασμούς, ε, και αυτή η χώρα είναι στον κλειό του Συμφώνου Σταθερότητας, τελικά ποιους βοηθάμε. Ε, αυτούς που τα πάνε καλά ή αυτούς που δεν έχουν σύγκληση ή που πλήττονται από κάποια σύμμετρο ε, κραδασμό. Άρα ε, δεν βλέπω τόσο πολύ να δίνεται προτεραιότητα σε αυτή τη σταθεροποιητική λειτουργία. Ποια είναι η απόψη για την πρόταση της Κομισιόν που υποτίθεται θα είναι η βάση για αυτή τη λειτουργία. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, ε, με τον συνεισηγητή μου, τον Ράιμερ Μπέγκ, έχουμε πει ότι καλό θα ήταν να υπάρξει διεύρυνση αυτής της υποστήριξη όχι μόνο για την προστασία των επενδύσεων, αλλά να υπάρχει και ένας μηχανισμός σε ό,τι αφορά ε, τις ε, παροχές ε, τις και συγκεκριμένα επιδόματα ενεργείας. Γιατί η γαλλογερμανική πρόταση δεν νομίζω ότι λαμβάνει υπόψη σε αυτή τη σταθεροποιητική. Thank Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στο ερώτημα που κάνατε για την κοινή δημοσιονομική ικανότητα. Το ότι συζητάμε το θέμα αυτό εκ νέου και με νέο ενθουσιασμό. Νομίζω ότι απαντά στο προηγούμενο ερώτημά σας σε ό,τι αφορά το θεματολόγιο ε, και αν είναι ρεαλιστικό. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια έχουμε προτάσεις από διάφορα φορείς, κράτη-μέλη, κομισιόν κτλ. Και αυτό από μόνο του είναι μια θετική ερθαρρυντική εξέλιξη. Φυσικά και είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση της Κομισιόν για αυτό το Ταμείο Σταθεροποίησης των Επενδύσεων όπως και άλλες προτάσεις ε, από τα κρατημέλη όμως. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Το πώς θα σχεδιαστεί αυτή η δημοσιονομική ικανότητα και το γεγονός ότι όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται τη σημασία του ζητήματος αυτού για την ίδια την επιβίωση της ΟΝΕ, την ύπαρξη της ΟΝΕ και αυτό από μόνο το είναι σημαντικό βήμα. Ο σχεδιασμό όμω δεν είναι κάτι εύκολο, του αντίον μάλιστα, για του λόγου ακριβώ που κι εσεί μα παρουσιάσατε. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, ότι αυτή η δημοσιονομική ικανότητα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε πρώτον να είναι επαρκή και ω προ το μέγεθο και ω προ το σχεδιασμό. Γιατί πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο ώστε να έχουμε αφενός πριν τον προκυκλικό χαρακτήρα παρά, ε, όπου θα γίνουν σεβαστοί κάποιοι κανόνες και μιλάμε για τους φυστάμενους κανόνες και θα το ξαναδούμε αυτό βέβαια τα επόμενα χρόνια Πρέπει να τηρούνται όμως κάποιοι κανόνες, όπως είπα, σε περίπτωση της κυκλικής ύφεσης. Αυτό μπορεί να είναι προκυκλικό. Και από την άλλη πλευρά, πρέπει να αντιμετωπιστεί και ο ηθικός κίνδυνος, ώστε να σχεδιαστεί δηλαδή ένας μηχανισμός που δεν θα ενθαρρύνει αποκλίνουσες συμπεριφορές. Ο σχεδιασμός λοιπόν της ικανότητας δεν είναι καθόλου απλός. Τι δείχνει η εμπειρία άλλων νομισματικών χώρων. Η τήρηση των κανόνων είναι θεμελιώδης κανόνες για τον συσκευασμένο προϋπολογισμό σε επίπεδο κράτου, σε άλλες χώρες και δικαιοδοσίες είναι θεμελιώδες επίσης ως αρχή. Επίσης όσο πιο αυτόματος είναι ο μηχανισμός τόσο καλύτερα λειτουργεί. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στις πολιτείες σταθεροποίηση ξεκινά από την καταβολή μικρότερου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει ύφεση επιβράδυνση Το δεύτερο είναι τα επιδόματα ανεργία. συγκέντρωση ε, των ε, μεταφορών εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη επίπτωση από την ε, κυκλική επιβράδυνση. Δεν θα γίνει μέσα σε μια μέρα ο μηχανισμός αυτός πρέπει να δούμε τι γίνεται σε άλλους ε, χώρους ε, νομισματικά ενοποιημένους. Δεν έχουμε ακόμα αυτή την ε, κατάσταση, άρα πρέπει να συνδυάσουμε το ρεαλισμό με τον οραματισμό στην προκειμένη περίπτωση. Είναι ό,τι και η πρόταση της Κομισιόν, ουσιαστικά ένα πρώτο βήμα. Σημαντικό φυσικά, πάρα πολύ σημαντικό που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και που κατατέθηκε αυτή η πρόταση. Αν δεν κανείς πώς ξεκινήσαμε, δεν γινόταν και πολλή συζήτηση παλαιότερα. Ήταν σαν να είχε εγκαταλειφθεί ως μη ρεαλιστικό, ως ανεδαφικό αυτό το ζήτημα. Με αυτό το έγγραφο πλέον σηματοδοτήθηκε η έναξη και δρομολογήθηκε αυτή η συζήτηση. Ραμόν Τρεμόσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Γκουαλτιέρη. Καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Θα κάνω δύο ερωτήσεις ε, στα αγγλικά. Το πρώτο ερώτημα νομίζω ότι είναι καλό ότι υπάρχει μεταξύ των Ευρωπαίων ρεκόρ αποδοχής για το ευρώ. Το νομισματικό μας σύστημα βασίζεται στην εμπιστοσύνη πολύ καλό το νέο αυτό. Ότι μετά από 20 χρόνια έχουμε τόσο μεγάλα ποσοστά αποδοχή για το ευρώ όμως, όπως ίσω γνωρίζετε σε ορισμένα κράτη-μέλη. Βλέπουμε ότι είναι δημοφιλής και η ιδέα ενός παράλληλου νομίσματος για την καταβολή επιδομάτων και για να ε, λυθούν τα προβλήματα και στον τομέα των δημόσιων δαπανών. Εγώ θεωρώ ότι είναι κακό το προηγούμενο αυτό, αλλά τέλος πάντων ε, θα ήθελα να απαντήσω και το δεύτερο ερώτημά μου αφορά την Ιταλία. Τη μόνη χώρα ουσιαστικά στην Ευρωζώνη που έχει καταφέρει πρωτογενές πλεόνασμα, νομίζω πριν από 19 χρόνια είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει ψηλό δημοσιοχρέος πολλά ε, πολλοί τόκοι πρέπει να καταβληθούν και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε αυτό το συνολικό ποσό του ετήσιου δημοσίου ελλείμματος. Εσείς πώς βλέπετε το ενδεχόμενο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός σταθερό να βοηθήσει την Ιταλία να αναχρηματοδοτήσει τα επιτόκια δημόσιου χρέους, να είναι δηλαδή κατώτερα, να είναι χαμηλότερα τα ποσά, χαμηλότερα επιτόκια, οπότε να διευκολυνθεί και η Ιταλική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Για το πρώτο ερώτημα μπορώ απλώς ε, να επαναλάβω την απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο παρελθόν. Το ευρώ είναι το μοναδικό νόμισμα της Νομισματικής Ένωσης. Επομένως, είτε αυτά τα παράλληλα νομίσματα είναι παράνομα, αν είναι νομίσματα δηλαδή όντως, δάλος δεν είναι νόμισμα και είναι χρέος και έτσι ε, προστίθενται στο υφιστάμενο χρέος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτη εναλλακτική εδώ. Για το δεύτερο ερώτημα, και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα ερωτήματα για την Ιταλία, να σας πω απλώς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει διάλογος. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να εξευρεθεί μια λύση και δεν νομίζω ότι τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να σχολιάσω αυτή την κατάσταση. Έχω πει πολλές φορές ότι οι υπερχρεωμένες χώρες θα πρέπει να περιορίσουν το χρέος τους, γιατί έτσι ενισχύουν ε, την ίδια τη θέση τους. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Πολύ σύντομα. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να μειωθεί το χρέος, ε, να μειώσουν μάλλον αυτές οι χώρες το χρέος τους. Αν δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, σχέση με πριν από 10 χρόνια, ίσως τώρα υπάρχει σε κάποια ε, κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη υπάρχει υψηλότερο δημόσιο χρέο. Έτσι έχουμε λιγότερα πολεμοφόδια για την αντιμετώπιση κάποια μελλοντικής κρίσης. Και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ ως έκτακτα μέτρα τα τελευταία χρόνια νομίζετε ότι πλέον μας θέτουν σε μια πιο αδύναμη θέση ή είναι επίγον για εμάς να περιορίσουμε το δημόσιο χρέος για να είμαστε πιο δυνατοί όταν έρθει μια επόμενη κρίση. Eh, eh, όταν το χρέος είναι πολύ ψηλό, αυτό αυξάνει την επάθεια μιας χώρας. Γίνεται πιο ευάλωτη, δηλαδή. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και νομίζω ότι το μάθημα ε, που άντλησαν πολλά, πολλές χώρες από την κρίση είναι ακριβώς αυτό, ότι όταν χτύπησε η κρίση δεν είχαν δημοσιονομικό περιθώριο παρέμβασης, γιατί ήταν υπερβολικά υψηλό το χρέος. Τώρα λοιπόν έχουμε ανάκαμψη που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, που συνοδεύεται από άνευ προηγουμένου χαμηλά επιτόκια. Και ε, οι διατάξεις της ε, πολιτικής μας θα πρέπει να αξιοποιηθούν για να ανοικοδομήσουμε αυτή την, ε, τη ζώνη ασφαλείας, αν θέλετε, για να είμαστε έτοιμοι την επόμενη φορά που θα υπάρξει μια κρίση και που θα χρειαστεί η κάθε κυβέρνηση να έχει στη διάθεσή της ένα τέτοιο δημοσιονομικό περιθώριο. Ευχαριστώ. Μόλις Σκοτ Κέιτο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο ασχολούμαστε με τις τρεις νομοθετικές προτάσεις για τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά που μας έστειλε η Οικονομισιόν. Όμως πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών για να χρηματοδοτηθεί το σύστημα. Χάρηκα που άκουσα στην ε, ομιλία του Μπενουά Κιουρέ αυτόν τον μήνα για την Κεντρική Τράπεζα και το Περιβάλλον ότι η ΕΚΤ εντός της εντολής της θα πρέπει να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα με δύο τρόπους. Πρώτον, ορίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού και δεύτερον, δρώντας αναλόγως, ε, ε, χωρίς βεβαίως να επηρεάζεται η σταθερότητα των τιμών. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς λίγα περισσότερα για το τι σημαίνει αυτό. Και οι συγκεκριμένες μου ερωτήσεις είναι πρώτον, μπορούμε να μας πείτε λίγα πράγματα για τα stress test σε σχέση με τον άνθρακα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, να έχει υποθεί ότι θα πρέπει να λαμβάνονται οι υπόψη εξωτερικότητες που ίσως προκαλέσουν χρηματοπιστωτική αστάθεια και κίνδυνη σχετική με το περιβάλλον. Οπότε, για να αντιμετωπιστούν υπερβαλλοντικοί συστημικοί κίνδυνοι θα θεωρήσετε πιθανόν να εισαχθούν πλαφών σε, στην επέκταση κάποιων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν το κλίμα και εμείς θα έπρεπε να υπάρχουν δεδομένη της σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης κάποια μέτρα που θα αφορούν ίσως την επιστοτική επέκταση συγκεκριμένων ρηπογόνων δραστηριοτήτων. Σας ευχαριστώ να πω πρώτα απ' όλα ότι συζητήσεις αυτές να σας δώσω τα γεγονότα. Κοιτάξαμε τις αγορές πράσινων ομολόγων, τα έσοδα από τα οποία χρησιμοποιούνται για επενδυτικά έργα με όφελος για το περιβάλλον. Και ο αντίκτυπος ε, που είχαν δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό μας δελτίο της 8ης Νοεμβρίου. Οπότε η ΕΚΤ έχει αγοράσει πράσινα ομόλογα και στο πλαίσιο αγορών στοιχείων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στο πρώτο σκέλος έχουμε αυτή τη στιγμή 24% του προγράμματος αγορών ε, των δημόσιο τομέα. επιλέξιμων ε, πράσινων ομολογών. Στο δεύτερο σκέλος ε, του ιδιωτικού τομέα έχουμε γύρω στο 20% και στα δύο προγράμματα το ποσοστό το οποίο έχουμε σε επιλέξιμα πράσινα ομόλογα αντικατοπτρίζει το ποσοστό σε ολόκληρο αυτό το σκέλος. Οπότε τα πράσινα ομόλογα είναι γύρω στο 4% των συνολικών επιλέξιμων στοιχείων. Οπότε τα στοιχεία δείχνουν ότι μέσω των αγορών αυτών το ευρωσύστημα έχει μειώσει τις ε, αποδόσεις πράσινων ομολόγων και στηρίξει την έκδοσή τους από μη χρηματοπιστωτικούς οίκους. Έχουμε και κάποιες οικονομετρικές αναλύσεις που αποδίδουν μεγάλο κομμάτι της πτώσης της ψαλίδας στα πράσινα ομόλογα στις δικές μας αγορές ε, ομολόγων του ε, εταιρικών ομολόγων. Κάτι το οποίο φαίνεται ιδιαίτερος μετά τις ανακοινώσεις μας ε, το Μάρτιο του 2016 και μετά την έναρξη του προγράμματος τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Ταυτόχρονα η έκδοση πράσινων ομολόγων αυξήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση και αυξάνεται έκτοτε. Και αυτό συμφωνεί και με προηγούμενα ευρήματα για τον αντίκτυπο στις αγορές εταιρικών ομολόγων. Τώρα, να απαντήσω στην δεύτερη ερώτησή σας. Οι προσπαθίες μας ε, Συγγνώμη. Ναι, οι κλιματικοί κίνδυνοι. Είχαν συζητηθεί και έχουμε καταβάλει κάποιες προσπάθειες που στόχο έχουν να στηρίξουν την, συμμετέχοντες στην αγορά, τους νομοθέτες και τους φόρους που ορίζουν προδιαγραφές για να καθοριστεί ένα σαφές πλαίσιο για να ανακατευθυνθούν οι χρηματοπιστωτικές ροές και να μειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί. Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης αυτής της πρόκλησης, η ΕΚΤ στηρίζει την δουλειά που γίνεται σε διεθνή φόρα και βρίσκεται και στο δίκτυο για το πρασίνισμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στο οποίο συνεργάζονται κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές ε, που στόχο έχουν να αναπτύξουν κοινέ πρακτικές για τα ζητήματα που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Να υπενθυμίσω ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ο μόνος δευτερεύον στόχος που έχει η ΕΚΤ. Σύμφωνα με τη συνθήκη θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να ερωτήσουμε γιατί να μην ε, προωθούμε βιομηχανίες που προωθούν την ανάπτυξη, όπως οι βιομηχανίες έντασης άνθρακα, ανεξαρτήτως οικολογικού αποτυπώματος. Εξίσου σημαντικό είναι το ότι η ΑΚΤ θα πρέπει να δρά σύμφωνα με τις αρχές μιας ε, ανοιχτής οικονομίας αγοράς ε, και του ανταγωνισμού. Και βέβαια η εντολή μας είναι να διασφαλίσουμε την σταθερότητα των τιμών. Ε, δηλαδή, κάνουμε ό,τι μπορούμε και οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε να επαναξετάζουμε το ζήτημα αλλά υπάρχουν και κάποια όρια στην έντολή μας εντός των οποίων πρέπει να κινηθούμε. Σας ευχαριστώ. Sorry, Marisa Matias, sorry. was not in this in the... Όχι λάθος, η Μαρίσα Ματίας είναι πρώτη. Ναι, Ρομπέρτο, δεν έφυγα, εδώ είμαι ακόμα. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε κύριε Τράκη που ήρθατε ξανά ενώπιον τη επιτροπή μας. Έχω τέσσερις ερωτήσεις. Οι δύο αρχικές αφορούν το ίδιο θέμα. Είπατε νωρίτερα ότι η κατάσταση της Ευρωζώνης όσο έχει αυτή τη στιγμή είναι κάτι προσωρινό. Εντός του 18 ήταν χαμηλά τα ποσοστά ανάπτυξης της Ευρωζώνης. Και το χαμηλότερο ποσοστό ήταν το τελευταίο τρίμηνο σε σχέση με τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Τι γίνεται με την ποσοτική χαλάρωση. Είχε αποφασιστικό ρόλο το μέτρο αυτό. Και ποια θα είναι η κατάληξη. Λέτε ότι θα λήξει σιγά σιγά το πρόγραμμα, αλλά με βάση τα δεδομένα που βλέπουμε έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Αν έχουμε τώρα πλήρη εξάρτηση της οικονομικής ανάπτυξης από μη συμβατική νομισματική πολιτική, μήπως είναι λάθος το μείγμα πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πω αλλιώς. Δεν φαίνεται τελικά μήπως ότι αν εξαρτώμεθα από μια ευνοϊκή για την ανάπτυξη νομισματική πολιτική και στα σχετικά μέτρα. Αν αυτό το συνδυάσουμε με πολύ χαμηλούς μισθούς και περικοπές, αυτό δεν πλήττει την ευημερία. Και είναι και μια ερώτηση που θέλω να κάνω και την έχουν πει και άλλοι, αλλά μήπως πρέπει πλέον να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, ώστε να αποδώσει το μέρο καλύτερα το μέτρο αυτό. Απάντηση. Θα απαντήσω αρχικά στο πρώτο ερώτημα. Στην εισαγωγική μου παρέμβαση μίλησα για την απώλεια αυτής της όθησης στην ανάπτυξη και αν είναι προσωρινός ή μόνιμος ο χαρακτήρας αυτής της επιβράδυνσης. Αυτή τη στιγμή, και γιατί λέω αυτή τη στιγμή, διότι θα συζητήσουμε όταν θα έχουμε το Δεκέμβρη τις τελευταίες προβολές αυτή ο πιο βραδύς ρυθμός, ε, η μικρότερη όφηση, έχει να κάνει πιο πολύ με την ε, εξομάλυνση της όλης διαδικασίας, ε, γιατί το 2017 ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Ε, υπό την έννοια ότι ήταν μια κατεξαίρεση κατάσταση. Έκτοτε η παγκόσμια ανάπτυξη και στα εμπορικά ζητήματα επιβραδύνθηκε σημαντικά και οι εξαγωγές επίσης. Υπήρξε λοιπόν αυτή η εξομάλυνση που εν μερή οφείλεται στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού που παρατηρούνται και σε άλλες συνιστώσεις και παραμέτρες που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη υπήρχαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως ε, για την αυτοκινητοβιομηχανία που μίλησα, αλλά και άλλοι προσωρινοί παράγοντες και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να εκτιμήσουμε τα δεδομένα και να πούμε ε, κατά πόσον αυτή η εικόνα είναι αυτό που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ή θα υπάρξουν αλλαγές. Αν μας περιμένει μπροστά σοβαρή ύφεση, μάλλον όχι. Αυτό θα ήταν η δική μου εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή πάντα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή σε ό,τι αφορά τι αγορέ, καθαρέ αγορέ περιουσιακών στοιχείων, μάλλον θα τι ολοκληρώσουμε φέτο. Και αν γίνει αυτό, η νομισματική πολιτική θα παραμείνει ευνοϊκή γιατί βασίζεται στην καθοδήγηση σε ό,τι αφορά τα επιτόκια και τις επανεπενδύσεις. Αυτά τα δύο συμπληρώνουν το ένα το άλλο και θα ενισχυθούν και στο μέλλον. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη στο δεύτερο ερώτημα δεν φαίνεται να συμφωνείτε ότι είχαμε πέντε χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, ότι είχαμε ανάκαμψη. 9,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί μέσα σε πέντε χρόνια. Δεν ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία της Ευρώπης τουλάχιστον. Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, ξέρετε σε διάφορα μέρη της Ένωσης βλέπουμε βελτίωση και ιδίως βέβαια σε όσες χώρες είχαν ψηλότερη δυνατότητα αξιοποίησης ε, και λιγότερες ελλείψεις εργατικού δυναμικού. σε άλλε χώρε όμω, και γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι ότι υπάρχει αυτή η σύγκληση και στα επιτόκια, είναι ότι οι δημοσιονομικέ πολιτικέ. Δεν βλέπω και τόσε περικοπέ στην Ευρωζώνη οι δημοσιονομικές πολιτικές, τουλάχιστον να δούμε τα σχέδια προπολογισμών σε όλες τις χώρες, με μία εξαίρεση, ε, σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, φαίνονται επεκτατικά αυτά τα σχέδια. Δηλαδή δημοσιονομικός προσανατολισμός είναι ουδέτερος προς ελαφρά ε, επεκτατικός. Τώρα, περισσότερη ευελιξία για προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Δύο παρατηρήσει από αυτού. Η δέσμη των νησιών των κανόνων ήδη δίνει κάποια ευελιξία για τα δημόσια προγράμματα επενδύσεων. Και το δεύτερο, αν ο κόσμο θέλει να το συζητήσουμε αυτό, αυτό σίγουρα είναι σημαντικό να συζητηθεί γιατί σε κάποιε χώρε υπάρχει σοβαρή έλλειψη υποδομών. Όμω, έχει γίνει εκτεταμένη και βαθιά συζήτηση η οποία γινόταν, ε, σχεδιαζόταν το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη και εκπονείται η συνδίκη του Μαστρίχτ. Δηλαδή ότι θα πρέπει οι δημοσιοπενδύσει να εξαιρούνται από τον ορισμό των δημοσιονομικών στόχων ή από τον προσδιορισμό των δημοσιονομικών στόχων. Η συλλογική απόφαση που ελήφθη τότε ήταν να μην εξαιρούνται από του ε, δημοσιονομικού στόχου. γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τι είναι δημόσια επένδυση και τι είναι τρέχουσα δαπάνη και μπορούμε να βρούμε πολλά παραδείγματα. Βέβαια, όλα είναι στα χέρια των νομοθετών. Εμείς κεντρική τράπεζα είμαστε, απλά. Thank you. Now, Γκέρολφ Θα μιλήσω Ολλανδικά, κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε για το τέλος ποσοτικής χαλάρωσης που είχε τελειώσει το 2015 κατ' ουσίαν μέσω της αγοράς αυτής ε, σχεδόν ενεργητικού δημιουργείται λεφτά. Με όλα αυτά για να διατηρηθεί σε λειτουργία ένα ασταθές ε, νομισμό τω μεταξύ βεβαίως ε, η νομισματική αυτή η πολιτική κατέληξε σε, μια, σε έναν έθισμο και υπάρχει ακριβώς ο κίνδυνος αυτός μετάβαση σε μια κανονική κατάσταση και βεβαίως ε, όλο αυτό οδήγησε σε καταστροφική κατάσταση. Είχαμε οντότες οι οποίες ε, διατηρήθηκαν στη ζωή χωρίς να έπρεπε και κράτη τα οποία δεν έκαναν πλέον προσπάθειες για να έχουν δημόσια, υγιή οικονομικά όπως το Βέλγιο το οποίο διόγκωσε τα προβλήματά του. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι έχουμε ανισορροπία στον τομέα των ε, ακινήτων και ολόκληρος ο χρηματοπιστωτικός ε, τομέας ουσιαστικά οδηγήθηκε προς τα εκεί γιατί η ποσοτική χαλάρωση σημαίνει ε, κατ' ουσίαν τεράστιες αγορές με φρέσκα ε, χρήματα και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια. Και βεβαίως φουσκώνουν πάρα πολύ οι ισολογισμοί των κεντρικών τραπεζών και έχουν φτάσει σε διατάσεις αεροστάτων. Λοιπόν, θα σταματήσει αυτό σε λίγες μέρες. Μας λέτε πως ε, υπό την αίρεση των δεδομένων ε, το ΔΣ υπολογίζει ότι θα σταματήσουν οι καθαρές ε, αγορές. Έχοντας λοιπόν υπόψη το πλαίσιο το οποίο ανέφερα και δεδομένου του εθισμού τον οποίο ανέφερα για κεντρικές τράπεζες και επιχειρήσεις Ποιου ε, κινδύνου βλέπετε μέσω μακροπρόθεσμα από το σταμάτημα και ποιες θανότητε να ξαναξεκινήσει η ποσοτική χαλάρωση. Thank you. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω σύντομα στο ερώτημά σα. Απλώ θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι η πολιτική μα είχε καταστροφικέ συνέπειες. Ναι. Δημιούργησε ναι 9,5 εκατομμύρια θέσει εργασία μέσα σε μερικά χρόνια. Η ανάκαμψη τη Ευρωζώνης σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην νομισματική πολιτική τη ΕΚΤ. Δεύτερον, αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ξαφνικά ε, να κινηθεί προ αυτήν την κατεύθυνση, όχι, δεν ήταν ξαφνική απόφαση, το είχαμε πει για τον Ιούνιο Καθόλου ξαφνική λοιπόν δεν είναι αυτή η απόφαση. Τρίτον, στο σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής για το σύνολο της Ευρωζώνης, όταν λέτε για το σύνολο, εννοείται όλες τις χώρες ε, χωρίς εξαιρέσεις και για όλους τους κλάδους. Δεν πρόκειται για μια νομισματική πολιτική ε, που στοχεύει σε συγκεκριμένους κλάδους, όπου κρατάμε τα επιτόκια χαμηλά ή υψηλά για κάποιον κλάδο αυτό θα γινόταν ή γινόταν στη Σοβιετική Ένωση, όχι σε μια ε, ευρωζώνη της ελεύθερης αγοράς. Ωστόσο, εκτιμούμε και θεωρούμε ότι και οι κυβερνήσεις αλλά και ε, ο ιδιωτικό τομέας και τραπεζικός και μη τραπεζικός ε, είναι έτοιμοι για μια τέτοια απόφαση σε περίπτωση που ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Να προσθέσω επίσης ότι η νομισματική πολιτική, ανεξάρτητα από την απόφασή μας για τις ε, καθαρές αγορές ε, στοιχείων ενεργητικού, θα συνεχίσει να ακολουθεί την ε, οδό που είχαμε μέχρι τώρα. Τα επιτόκια δηλαδή δεν θα αυξηθούν μέχρι μετά το καλοκαίρι, λέγαμε, στο EIS της ΕΚΤ. E και μετά λέμε ότι η ΕΚ θα επανεπενδύσει τα ομόλογα ε, που θα οριμάσουν για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Thank you, Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάγκε. Αντίθεση με τον προλύσαντα, εγώ θεωρώ ότι μπορείτε μετά από 7 χρόνια να κοιτάξετε το παρελθόν και να αισθάνεστε επιτυχής γιατί χωρίς παρεμβάσεις σας δεν θα ήταν τόσο σταθερό το ευρώ και αν γιορτάζουμε τα 20 χρόνια αυτό οφείλεται στην ΕΚΤ παρά την κριτική που έχουμε για την πολιτική των επιτοκίων και το πρόγραμμα των αγορών θεωρώ ότι η δουλειά σας είναι σημαντική. Τώρα όμως έχουμε νέες προκλήσεις. Έχω τρεις ερωτήσεις. Το πρώτο είναι ο πληθωρισμός. Είπατε ότι ο βασικός πληθωρισμός είναι χαμηλός, ο συνολικός είναι κάπως υψηλότερος, περιλαμβάνει και την ενέργεια που έχουμε ξεπεράσει το 2% και που απαιτούνται μέτρα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την ε, σύγκληση. Οι νέες έρευνες δείχνουν πως όλες οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν ε, θετική σύγκληση με την εξαίρεση της Ιταλίας, η οποία όμως έχει και άλλες δυσκολίες γιατί η δημόσια η πρόσφορά σας για 220 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το 1 τρίτο πήγε στην Ιταλία και έχουμε βεβαίω και τις πολιτικές εξελίξεις που οδηγούν σε πόλη σε κρατικών ομολόγων. Είναι σε θέση η ΕΚΤ να δώσει άλλη μια ένεση ρευστότητα στις Ιταλικές τράπεζες όπως διάβασα σήμερα στις εφημερίδες. Και τρίτον, το τρίτο αφορά την αισιοδοξία σας ότι υπάρχει ένα αποτελεσματικό ή ότι θα έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα συντονισμού της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Η πείρα των τελευταίων 20 ετών αμφισβητεί κάτι τέτοιο. Και μετά μιλήσατε για την μετάβαση από τον συντονισμό στην ε, κοινή λήψη αποφάσεων, η οποία βεβαίω είναι μια αργή διαδικασία, μα περιμένουμε ήδη αρκετά χρόνια πότε βλέπετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον μελλοντικό μηχανισμό σταθερότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέσατε πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια στην αρχή της παρέμβασής σας. Αρχικά, λοιπόν, για τον πληθωρισμό. Ε, φυσικά και ο headline inflation είναι αυτός που μας ενδιαφέρει εμάς. Ε, τώρα ο πληθωρισμός αυξάνεται τελευταία εξαιτίας ε, των τιμών και του κόστους ενέργειας. Και οι ενεργικές τιμές όμως θα πέσουν, οπότε αναμένεται και πτώση αυτού του πληθωρισμού στους επόμενους μήνες και αυτός ο πληθωρισμός λοιπόν. Όμως ε, και τα αστικά στοιχεία αυτού του πληθωρισμού είναι πιο σταθερά από ό,τι ενέργεια και άλλα στοιχεία. Γι' αυτό και το αποκαλούμε ε, βασικό πληθωρισμό, ε, ο οποίος όπως είπα εισαγωγικά έχει κάπως μετριαστεί, είναι μικρός ο πληθωρισμός, <clears throat> αλλά χαμηλότερο, υψηλότερος από ό,τι στο παρελθόν τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο βασικός πληθωρισμός θα αυξηθεί. Οι ονομαστικοί μισθοί που αυξάνονται σε ορισμένες χώρες περισσότερο από τις άλλες. Όμως είναι σίγουρα ποιοτικά καλύτερη αυτή η αύξηση των μισθών σε σχέση με το παρελθόν. Στο παρελθόν είχαμε μία προσωρινή μόνο αύξηση των μισθών που οφειλόταν ε, σε κάποιον συγκεκριμένο παράγοντα. Τώρα όμως έχουμε να κάνουμε με μισθούς που προκύπτουν μετά από διαπραγματεύσεις. Πρόκειται λοιπόν για μια σταθερή αύξηση που ε, θα είναι μακροχρόνια. Σταδιακά αυτές οι μισθολογικές αυξήσεις και παράλληλα και των ε, τιμών των καταναλωτών θα περάσουν ε, σε υψηλότερες τιμές και σε υψηλότερο πληθωρισμό στο μέλλον. Αυτό, ανάλογα με τη χώρα, θα εξαρτηθεί και από το στάδιο του οικονομικού επιχειρηματικού κύκλου. Συνήθως βλέπουμε ότι στην αρχή αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, αλλά η ποιότητά τους είναι κακή. Είναι προσωρινές θέσεις εργασίας. Και όταν κάποιο έχει μια προσωρινή θέση εργασία, δεν διεκδικεί και αύξηση μισθού. Σταδιακά σταθεροποιείται η θέση τους και μετά ζητούν ε, υψηλότερο μισθό. Αυτό είναι ο συνήθι κύκλο. Κάποιε χώρε είναι πολύ προηγμένε. Ε, Συνήθω οι θέσει απασχόλησης είναι μόνιμες. Ενώ σε άλλες χώρες ο μεγάλος όγκος των θέσεων εργασίας παραμένει ε, προσωρινός. Γενικά όμως το μερίδιο των ε, καλών θέσεων εργασίας αυξάνεται, γι' αυτό θα δούμε ότι θα οριμάσει η αγορά εργασία. Αυτοί οι δύο παράγοντες λοιπόν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αυξήσει θα ε, μεταφραστούν και σε υψηλότερες ε, τιμές. Όμως όλα αυτά παίρνουν χρόνο γιατί για πολύ μεγάλο διάστημα δεν υπήρχαν επαραίτητες συνθήκες για να φτάσουμε εδώ. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχει σύγκληση του πληθωρισμού προς του στόχους μας. Μιλώντας για σύγκληση, συμφωνώ απολύτως. Και να σας πω και το εξής. Σας μίλησα για έκανα μια μνήα σε αυτή την, σε ατζέντα από την μετακίνηση ε, προς τους θεσμούς αντί για τους κανόνες. Όμως για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται εμπιστοσύνη μεταξύ των ε, χωρών μελών, μεταξύ των κυβερνήσεων, μεταξύ των λαών. Και όλα αυτά εξαρτώνται από δύο στοιχεία. Ο σεβασμός και τήρηση των κανόνων και δεύτερον αυτό που αναφέρατε, η σύγκληση. Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει απόκληση μεταξύ των χωρών, ε, αυτό οδηγεί σε εγγενή αδυναμία τους. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να τους εμπιστευτεί κανείς σε μια διαδικασία που εμείς θεωρούμε αναπόφευκτη για μια ισχυρή νομισματική ένωση. Κάτι τελευταίο για την μετάβαση αυτή προς τη σύγκληση με βάση τους θεσμούς και όχι με βάση τους κανόνες. Δείτε τι γίνεται με την νομισματική πολιτική. Μέχρι τα τέλη τη δεκαετία του 80 κάθε κεντρική τράπεζα έχει δική της νομισματική πολιτική. Και από πλευράς ε, χρηματοοικονομικής ε, σταθερότητα τη κάθε τράπεζας ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί είχαμε ελεύθερη σκηνή κεφαλαίων, αλλαγέ ε, των ισοτιμιών συνεχώ και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να χειριστεί κανεί την κατάσταση. Και τότε μάλιστα υπήρχαν κανόνες σταθεροποίησης ε, των ισοτιμιών, κανόνες που ρύθμιζαν ε, ε, το εύρος κίνησης των συναλλαγμάτων. Όλα αυτά όμως παραβιάζονταν συνεχώς γιατί υπήρχαν πολύ ισχυρές πιέσεις της αγοράς έτσι οδηγηθήκαμε στην σύσταση της ΕΚΤ και αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα της μετάβασης ε, από τη σύγκληση με βάση τους κανόνες, τη σύγκληση με βάση τους θεσμούς και βάσει και με αυτά που είπατε και εσείς, η μετάβαση ήταν εξαιρετικά επιτυχής. Σας ευχαριστώ. Πέντρο Σίλβα Περέιρα, παρακαλώ. Yeah. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Ντράγκη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω τα βασικά μηνύματα που μας απευθύνατε σήμερα. Πρώτον, ότι απαιτείται ακόμα σημαντική παροχή ε, νομισματικών κινήτρων που θα διατηρηθεί και μετά το τέλος των ε, καθαρών αγορών ε, στοιχείων ενεργητικού και ότι η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας καθιστά αυτή την κίνηση κατανοητή και ότι απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα προς τη μεταρρύθμιση ναι. Μιλήσατε για τον συντονισμό πολιτικής, την θέσπιση μιας ε, λειτουργίας θεραπείας επενδύσεων και ε, της AICM. Έχω τα εξή ερωτήματα. Πρώτον, για την λειτουργία θεροποίηση. Είπατε ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται αυτή την λειτουργία για να διατηρήσει τη σύγκληση. Συνήθως ε, είστε μετρημένος στα λόγια σας. Θεωρείτε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη σύγκληση και όχι ε, να την προωθήσουμε περαιτέρω. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε κατάσταση απόκλησης και από οικονομικούς και, και με βάση τους κοινωνικούς όρους στα μέλη της Ευρωζώνης. Δεύτερον, για τη μεταρρύθμιση ASM ε προβλέπεται η θέσπιση του ενιαίου Ταμείου Εξεγίενσης. Ε, πόσο επίγει όμως αυτό το ζήτημα. Γιατί κάποιοι λένε ότι πρέπει ε, να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα όπου θα καταστεί πλήρως λειτουργικό αυτό το ταμείο. Και σήμερα η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα εξετάσει την έκθεσή μου για τη μεταρρύθμιση και θεωρούμε ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παρακολούθησης θα πρέπει νομισματικό ταμείο θα πρέπει να γίνει Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας. Ποια είναι η δική σας νόμη. Thank you. Ευχαριστώ. Οι λέξει ε, να διατηρηθεί η σύγκληση αναφέρονται σε μια κατάσταση όπου οι χώρες έχουν συγκλίνει αρκετά για να έχουν μια κεντρική δημοσιονομική ικανότητα αλλά εξακολουθούν να υφίστανται καρατασμούς ε, ιδιαίτερους ή διαφορετικών, όπου η διαφορετικων οπου η συγκληση θα χαθεί εάν δεν ε, γίνει κάτι. Με αυτήν την έννοια χρησιμοποιείται η λέξη να διατηρηθεί η σύγκληση. Το ενίο ταμείο αυτό διάσωσης είναι κατεπήγον και ακριβώς ε, είναι ένας από τους εύκολους στόχους όπως λέμε στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί και αποφασιστεί και έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες ακόμα. Πρόκειται λοιπόν για κατεπήγοντα μέτρα και αυτό είναι μέρος της ε, εμβάθυνσης ε, και του να γίνει η νομισματική ένωση ισχυρότερη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση, να προχωρήσουμε μπροστά με τρόπο αξιόπιστο στην ένωση κεφαλαίου αγορών. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα και γρήγορα. Αλλά θα χρειαστούν καιρό, παραδείγματο χάρη, ο αναρμονισμός ε, της νομοθεσίας περί χρεοκοπίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα και πιστεύω ότι η Κομισιόν προσεχώς θα συντάξει ένα έγγραφο όπου θα ορίσει τους εύκολους στόχους της Ένωσης Κεφαλαίων Τρίτων. Ε, δεν πράγματι διαφωνώ καθόλου μαζί σας, ε, συμφωνώ πλήρως ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λέξη νομισματικός ε, για το νέο αυτό θεσμικό όργανο. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, βεβαίως. Πράγματι. Είναι κάτι το... Πάρα πολύ καλό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας, λέει ο Πρόεδρος, και πολύ που μας το στηρίζουμε. Ευχαριστώ, κύριο Νίντερμαϊρ. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι Συμφωνώ και με την αξιολόγηση του κυρίου Λάγκεν για την ε, πολύ καλή δουλειά που κάνατε στην ΕΚΤ. Έχω μία ερώτηση για τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, αλλά όπως είπατε η οικονομία αυξάνεται, ε, ωφελείται από τη μείωση της ανεργίας και αυτό οδηγεί σε περαιτέρω οικονομική επέκταση γιατί περισσότερος κόσμος έχει ε, δουλειά και άρα έχει και περισσότερο εισόδημα. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουμε και ανάπτυξη. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσει έχοντας κατά νου τα τελευταία στοιχεία που δεν είναι ιδιαίτερο ισχυρά. Η πρώτη είναι ότι εάν υπάρχει κάποια ορατή επιβράδυνση τα επόμενα ένα-δύο χρόνια έχουμε επαρκή εργαλεία για να στηρίξουμε την οικονομία. Η ανησυχία μου είναι και το είπατε κύριε Πρόεδρε πως η δημοσιονομική πολιτική είναι επεκτατική αυτή τη στιγμή τα επιτόκια είναι γύρω στο μηδέν Μας δείπουν λοιπόν δύο στοιχεία για να σταθεροποιήσουμε την ανάπτυξη αν επιβραδύνει η οικονομία. Και δεύτερον, ένα άλλο ζητήματα, είπατε ότι η αυτοκινητομηχανία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στα στοιχεία του τριτού τριμήνου. Αλλά έχουν εντύπωση ότι τα εργοστάσια παράγουν τα αυτοκίνητα, απλά δεν γίνονται οι πωλήσει γιατί δεν υπάρχουν εγκρίσει τύπου, αλλά υποθέτω ότι ε, περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ ε, εάν υπάρχουν τα αυτοκίνητα εκεί και δεν υπάρχει η προσθέμενη αξία της πώληση. Αναρωτιέμαι λοιπόν σε ποιο βαθμό μπορεί η αυτοκινητοβιομηχανία να εξηγήσει την ανεμική ανάπτυξη του ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο, ειδικά στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση. Αν υπάρχει ορατή επιβράβευση τα επόμενα έτη. Θα έχουμε αρκετό χώρο για άσκηση πολιτικής. Η απάντηση είναι ότι η νομισματική πολιτική που ασκούμε θα παραμείνει ε, πάρα πολύ υποβοηθητική. Ακόμη και για παρατεταμένη χρονική περίοδο διότι τη σύγκληση του πληθωρισμού στο στόχο μας βλέπουμε να έχει ένα ορίζοντα 2020 με βάση τις εκτιμήσεις μας. Και αυτό το βλέπουμε και από τα επιτόκια και από το, την πολιτική που εφαρμόζουμε, την επενδυτική κτλ. Σε ό,τι αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, υπάρχει αυτό το τρίμηνο βελτίωση, όχι στον βαθμό όμως που να τη σταθμίζει την υποχώρηση του προηγούμενου τριμήνου. Ίσως χρειαστεί πάνω από ένα τρίμηνο για να δούμε ακριβώς ε, να αντισταθμίζεται αυτή η κατάσταση. Αλλά δεν βλέπουμε λόγους να μην υπάρξει ανάκαμψη. Απλά θα σας δώσω και μια προειδοποίηση στη συνέχεια. Ε, δεν είναι όμως μόνο εκεί ασθενέστερη η ανάπτυξη. Υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες για την αυτοκινητομία και άλλοι που επηρεάζουν. Χαμηλότερο απτυξιακό δυναμικό, και λόγω των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών. Γιατί λέμε ότι πρόκειται για επιβράδυνση. Γιατί η παγκόσμια εμπορική ανάπτυξη είναι με χαμηλότερη αλλά χαμηλή. Έχουμε δει χαμηλότερου δείκτε εμπιστοσύνη που είναι πάνω όμω από τι ιστορικά, τις ιστορικές μέσα στη μέσα. Ίσως και ρεκόρ για κάποιες εποχές. Άρα αυτή τη στιγμή είναι ακόμα πρόωρο. Το είπα και πριν, θα έχουμε σύντομα νέα στοιχεία. Είναι πρόημο, πρόωρο να πει κανείς ότι έχουμε επιβράδυνση. Και είπα ότι υπήρχαν κάποιοι παράγοντες και στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλες χώρες. Γιάκοπ Φον Βάιτσέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τράιτ. θα συμφωνήσω με τους Νίτερ Μάγερ και Λάγκεν ε, στην ε, συνολικά αισιόδοξη εκτίμηση της κατάστασης ε, και με χαρά θα το κάνω. Επίσης μας δώσατε κάποιες έτσι κλεπτισμένες εξηγήσει όταν ο ήλιος καίει καλό είναι να φτιάξουμε την οροφή για να είναι στεγανή όταν αρχίσουν οι βροχές. Κάτι τέτοιο νομίζω είπατε λίγο πολύ. Να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη καταιγίδα, αλλά βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις ε, των χωρών με πολύ υψηλά ε, επίπεδα χρέους και πολύ χαμηλά ποσοστά ανάπτυξη. Άρα ο ήλιος μπορεί να καίει και πολύ πριν βρέξει. Το θέμα είναι πώς θα ενισχύσουμε την νοσονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Αυτό είναι σημαντικό συστατικό για να επισκευάσουμε τη στέγη, αν θέλετε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και επειδή μιλήσατε για τη σύγκληση, τη χρησιμοποίησατε τη λέξη αυτή στην ομιλία σας. Παραδοσιακά νομίζω θα σκεφτόταν κανείς ότι η έννοια σύγκληση σε αυτό το πλαίσιο είναι κάτι παραγωγικό και χρήσιμο γιατί μπορεί να περιλαμβάνει κάτι που στις Βρυξέλλες αρεσκόμαθε να το αποκαλούμε δημιουργική ασάφεια. Όλοι θέλουν να ακούνε αυτό που τους αρέσει να ακούνε, αλλά εγώ φοβάμαι κάπως. Αυτή η λέξη, σύγκληση ως ασαφής και αόριστη, έχει γίνει ως ένα βαθμό πρόβλημα. Διότι δηλαδή υπάρχει φυσικά η λέξη σύγκληση. Τα κράτη-μέλη που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ελλαγματικές ισοτιμίες ή άλλους μηχανισμούς και έχουν μικρό δημοσιονομικό περιθώριο, μπορούν έτσι να αντιμετωπίσουν τους κραδασμούς. Είναι ένα είδος εξασφάλισης, ε, προετοιμασία αντιμετώπισης ε, κραδασμών. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος σύγκλησης επίπεδο. Όπου εδώ έχουμε τα διαρθωτικά ταμεία. για να ενθαρρύνουμε τη συνολική οικονομική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν κατανάγει κάτι που είναι ίδιον τη νομισματική πολιτική και πρέπει να σα πω ότι σε κάποιε χώρε, σαν η σύγκληση θεωρείται ε, ή αντιμετωπίζεται ε, από την ευρεία της αυτή έννοια. Μιλάμε για μια ένωση μεταφορών πιστώσεων σε μεγάλο βαθμό. Θα ήταν πιο λογικό ίσως, έτσι θεωρώ εγώ, να αποχαιρετήσουμε όχι το στόχο της Εκκλησίας, αλλά την χρήση της έννοιας αυτής σε αυτό το πλαίσιο για να επιχειρηματολογούμε βάση αυτής για τη δημοσιονομική ικανότητα στην Ευρωζώνη. Και είναι ίσως έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο γρήγορη πολιτική συνένεση για το τι χρειαζόμαστε. Παραδείγματο χάρη αυτή η επανασφάλιση κατά της ανεργίας. Και κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις σε σχέση με το τι εννοούμε και με τον ευρωπαϊκό τα κτλ. I completely Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Την ώρα που μιλούσατε σκεφτόμουν τι είδους σύγκληση τελικά εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Και υπάρχουν τουλάχιστον τρία διαφορετικά είδη σύγκλησης. Τρία φαινόμενα ουσιαστικά περιγράφει. Κυκλική σύγκληση καταρχάς. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Η σύγκληση ως ποσοστό ανάπτυξης. Υπάρχει και αυτός ο δείκτης διασποράς που βλέπει την προσθέμενη αξία της ανάπτυξης. Αυτός ο δείκτης σήμερα είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αρχές της δεκαετίας του 90 πρέπει να τρέξουμε για να βρούμε αντίστοιχα χαμηλά ποσοστά, άρα η σύγκληση έχει γίνει, υπ' αυτή την έννοια, λόγω της ανάκαμψης κυρίως. Πριν, με την κρίση υπήρχε μεγάλη απόκληση. Δεύτερη σορισμός της σύγκλησης. Διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Με αυτό συνδέεται. ουσιαστικά η σύγκληση που πρέπει να έχουμε. Αυτή είναι. Ένα παράδειγμα. Αναφέρατε και συμφωνώ μαζί σας. Αυτό το σχέδιο επιδόμηση ανεργία η ασφάλιση ανεργία είναι ελπιδοφόρο μονοπάτι. Αλλά οι αγορές εργασία διαφέρουν. Οι κανόνες ταξινόμηση δεν διαφέρουν ε, εντελώς. κάποιοι ορίζουν ένα κεντρικό επίπεδο, αλλά κάποιοι άλλοι όχι. Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση λοιπόν. Πρέπει να έχουμε σύγκληση θεσμών επί ή πραγματικών διαφορετικών μεταρρυθμίσεων ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική οικονομία και να υπάρχει σύγκληση και σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Γιατί αν έχουμε μια πολύ ανταγωνιστική οικονομία και μια καθόλου ανταγωνιστική οικονομία, είναι πολύ δύσκολο αυτέ οι οικονομίες να κάνουν κάτι από εκείνο. Και έχουμε και τον τρίτο, την τρίτη έννοια σύγκληση, αυτό που είπατε για τα καταμία. ταμεία. Δηλαδή, αναδιανεμητική σύγκληση. Σύγκληση που επιτυχάνεται δια τη αναδιανόμηση. Νομίζω ότι ο πρώτος ορισμός είναι αυτός που πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε. Έναντι δηλαδή αφόρων φάσεων, αφόρων κραδασμών. Οπότε καλό θα ήταν ίσω πράγματι να χρησιμοποιούμε καθόλου την έννοια αυτή, τον όρο σύγκληση δηλαδή. Ευχαριστώ. το σκεφτούμε, θα το σκεφτούμε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς εδώ εξετάζουμε τους ασύμετρους κρατασμούς, οπότε είναι σαφές ότι πρόκειται για το πρώτο είδος ε, σύγκλησης. Ουσιαστικά αυτό για την ανασφάλιση ανεργίας είναι ένα μέτρο έκτακτης ανάγκης που αφήνουν ένα περιθώριο λιγμών στα εθνικά συστήματα. Εντάξει, και το τρίτο είδος σύγκλησης διαφέρει, αλλά και αυτό είναι σημαντικό και απαραίτητο. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό γιατί αφορά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από σημαντική άψη είναι σημαντική αυτή η διάκριση. Περβόνς, έχεις το λόγο. Ο κύριος Λούκε δεν είναι εδώ. Yes, but, uh, but uh, if you, Sorry, that's. Otherwise, we, we, we start with Philip and then you, you, okay. Ο Φίλιπ, λοιπόν. Φίλιπ Λάμπερτς. Ευχαριστώ, είναι πάντα χαρά να σας έχουμε εδώ. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε πριν για το πώς θα περάσουμε σε ένα σύστημα με βάση τα θερμικά όργανα και όχι με βάση τους κανόνες. Θα ήθελα να ακολουθήσω το σκεπτικό της συναδέλφου μόλις Κοτ Κέιτο, γιατί άκουσα μεγάλη προσοχή την απάντησή σας και Μπορώ να σα πω ότι δεν με καλύψατε πλήρω, γιατί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλαπλοί περιορισμοί και στόχοι. Μπορεί να θέλουμε να συνεχίσουμε να ε, ε, χρηματοδοτούμε δραστηριότητες ε, που είναι θετικές για την απασχόληση, πολύ αρνητικέ όμως για το κλίμα. Αλλά τελικά, αν αφήσουμε την κλιματική αλλαγή να ολοκληρωθεί, δεν θα υπάρχει οικονομία πια. Τι θέλω να πω, πράγματι, στο πλαίσιο της προσθετικής χαλάρωσης, η ΕΚΤ και των δραστηριοτήτων της, η ΕΚΤ χρηματοδοτεί δραστηριότητες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση ή το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Όμως, εξακολουθεί να χρηματοδοτεί δραστηριότητες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και αυτό είναι που με προβληματίζει, γιατί αν δείτε τη δυναμική της αγοράς, λέτε ότι εμεί είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς με απόλυτη προσήλωση. Ναι. Όμως αυτή η βραχυπρόθεσμη αιμονή με την ε, ελεύθερη αγορά δεν λαμβάνει υπόψη ε, την κλιματική αλλαγή σε ό,τι αφορά την λήψη αποφάσεων. Και σε αυτή την περίπτωση, αν ισχύει αυτό δηλαδή, τότε θα έχουμε μια δυναμία της αγοράς. Και αφενός έχουμε λοιπόν τα όσα κάνει η ΕΚΤ με τα μέσα της ε, και αφετέρου έχουμε τις δικές μας δυνατότητες να ρυθμίσουμε την οικονομία. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένας μηχανισμός δεσμευτικής ρήτρας για να υπάρχει κάποια πειθαρχία στην ε, αγορά. Θα ήθελα και τις δικές σας σκέψεις προς αυτό, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας ε, του συστήματος εποπτείας. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν αποσυνδέουμε τον ε, την ανάπτυξη από τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ε, πώς ε, λύνονται όλα αυτά. Ναι, δεν είναι εύκολο. Ναι, δεν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε ε, και σκεμμένα, δηλαδή δεν χρηματοδοτούμε δραστηριότητες που αυξάνουν την απασχόληση και ζημιώνουν το περιβάλλον. Ανέφερα όλες ε, τις ε, δευτερεύουσες αρμοδιότητες ε, της ΕΚΤ. Έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση στο Συμβούλιο και προτίθεμαι να τη συνεχίσω. Πώς μπορούμε δηλαδή, εάν μπορούμε, να επεξεργαστούμε περαιτέρω την οικονομική μας πολιτική. Για το χαρτοφυλάκιο των συντάξεων, των συνταξιωτικών ταμείων, έχουμε στραφεί προς ε, μάνατζερ που έχουν ε, προσυπογράψει συγκεκριμένε ε, αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και, και, απαιτείται από εκείνου να λαμβάνουν υπόψη και συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά πρότυπα στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, εξετάζουμε το δεχόμενο να διευρύνουμε τις δυνατότητες του επιτελείου μας να επενδύουν και σε βιώσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουμε ξεκινήσει και μία εσωτερική ε, έρευνα για το πώς ε, τα κριτήρια του ΟΗΕ θα μπορούσαν ε, να υλοποιηθούν και στη δική μας δραστηριότητα. Προσπαθούμε λοιπόν, δεν είναι εύκολο, γιατί η νομισματική πολιτική αφορά ολόκληρη την Ευρωζώνη, όλες τις χώρες, όλους τους κλάδους. Ενώ οι στόχοι μας προσδιορίζονται σορευτικά. Όμως, Όλο ένα και περισσότερο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ε, ασχολούνται και προβληματίζονται για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. κυρία Μπαγάς. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. σχεδιάζετε την ε, επιστροφή προς ε, τα συμβατικά ε, μέσα άσκησης νομισματικής πολιτικής που επεσήμανε και ο συνάδελφος Σίλβα Περέιρα. Όμως, πέραν τούτου, και ένα ερώτημα που ήδη σας έχω θέσει, αλλά το θέτω εκ νέου, για, την, για το στόχο ότι αφορά τη σταθερότητα των τιμών δίνεται μεγάλη έμφαση ε, στις ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, τα αναφέρεται συχνά, όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που, όπου, οδηγούν ε, στο συμπέρασμα ότι δεν θα αυξηθεί αρκετά η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είτε αυτό έχει να κάνει με δημογραφικούς, δημογραφικές αιτίες, είτε με την παραγωγικότητα στα κράτη-μέλη. Όταν όμως επιστρέψετε ε, στη συνηθισμένη λειτουργία σας, ο στόχος του 2% θα είναι πάντα ο στόχος που θα έχετε για τον πληθωρισμό. Um, Ευχαριστώ. Το είπα νομίζω και πριν ότι αυτή την στιγμή είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε με σιγουριά το εάν μέσω μακροπρόθεσμα να βρισκόμαστε σε μια πορεία στάσιμότητας όπως λέγεται ή εάν υπήρχε απλά μια προσωρινή πτώση της ε, ανάπτυξης. Γεγονός είναι ότι αυτό το οποίο είδαμε τα τελευταία 6-7 χρόνια είναι ότι οι δυνατότητες ε, ανάπτυξης ανέκαμψαν Οπότε δεν σημαίνει ότι ε, θα παραμείνουν πάντα σε αυτό το χαμηλό επίπεδο. Βεβαίω υπάρχουν και παραγόντε που αναφέρονται όπως η δημογραφία, αλλά από την άλλη έχουμε και την ψηφιοποίηση. Έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις ε, παντού που από την άλλη θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να καταστήσουν λιγότερο πιθανή την ε, στασιμότητα αυτήν. Είναι πάρα πολύ ευεβαιω κάτι τέτοιο αυτήν την στιγμή. Και έτσι θα έλεγα καθορίζουμε και την νομισματική μας πολιτική εξαρτάται από την σύγκληση την ε, μόνιμη μέσω σύγκληση. Και στο πλαίσιο αυτό ρωτάτε αν το 2% εξακολουθεί να είναι στόχο. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι πολλοί μου έκαναν αυτή την ερώτηση υπονοώντα ότι θα πρέπει να έχουμε 1% ή 3%. Και η απάντηση πάντα είναι ότι δεν ε, είναι τυχαία που επέλεξαν όλες οι κεντρικές τράπεζες ε, σε ολόκληρο τον κόσμο στα τέλη της δεκαετίας του 90 το 2%. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, είναι πάρα πολύ σημαντικοί σε μια νομισματική ζώνη όπου δεν ε, συμβαίνουν τόσο συχνά αυτές οι αλλαγές συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οπότε ο περιορισμός σε ένα χαμηλότερο επίπεδο πληθωρισμού θα κάνουν αυτές τις προσαρμογές πιο δύσκολες από ό,τι θα ήταν με ένα υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού. Επίσης, είναι δύσκολο να πούμε ότι αλλάζουμε έναν στόχο αυτή τη στιγμή τον φτάσουμε. Δεν θα ήταν αξιόπιστο αυτή την στιγμή, αλλά βεβαίω υπάρχουν λόγοι για τους οποίους δεν συζητάμε μια τέτοια επιλογή, γιατί οπωσδήποτε μπορεί να αυξηθεί, να αυξηθούν οι αναταράξεις και να επηρεαστούν οι προσδοκίε. Οπότε για την ώρα θέλουμε να προχωρήσουμε και ειλικρινά μέχρι στιγμή δεν σκεφτόμαστε κάποια αλλαγή στου ε, στόχους. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε τελειώνουμε με το πρώτο μέρος του νομισματικού διαλόγου με τον κύριο Ντράγκη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας και θα ήθελα νομίζω να υπογραμμίσω την ευρύτατη στήριξη της νομισματικής σας πολιτικής από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα που προέκυψε σήμερα και να παραλάβουμε τη σημασία αυτού του διπλού μηνύματος που δώσατε που όπως είπαμε ε, το στηρίζω και εγώ και τώρα περνάμε στην ακρόαση με τον Μάριο Ντράγκη υπό την ιδιότητά του ως ε, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας που όπως ξέρετε είναι αρμόδιος φορέας για την μακροπροληπτική εποπτεία του συστήματος και τελευταία φορά είχε έρθει υπ' αυτήν την ιδιότητα ο κύριος Ντράγκη στις 9 Ιουλίου 2017 2018 νομίζω 18 νομίζω. Και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το Κοινοβούλιο εργάζεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΣΕΖΑ. Οπότε καλώς ήρθατε υπ' αυτήν την ιδιότητα και έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ τη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κυρίε και κύριοι, με μεγάλη χαρά Απευθύνομαι σε εσά για δεύτερη φορά απόψε. Αυτή τη φορά από την ιδιότητά μου ω πρόεδρο ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Θα ήθελα να εστιάζω σήμερα σε δύο θέματα. Πρώτα θα σα αναφέρω κάποια από τα πορίσματα του έργου του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σε ό,τι αφορά τα εμπορικά κίνητα και έπειτα θα σα ε, αναφέρω τι προτάσει του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα μακροπροληπτικά εργαλεία για τους ασφαλιστές. Καταρχάς, εμπορικά κίνητα. Πρόκειται για έναν τομέα σημαντικό για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όχι λόγω των διαστάσεων που έχει, αλλά και επειδή είναι στενά συνδεδεμένος με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και άλλα τμήματα της πραγματικής οικονομίας. Γι' αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό οι αρχές μακροπροληπτικής εποπτείας να παρακολουθούν εκ του σύνοικης της εξελίξης στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Σήμερα το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου δημοσιοποιεί τα πορίσματα της ε, παρακολούθησης του τομέα. Και θέλω να σας ε, παρουσιάσω ορισμένα τα βασικά θέματα αυτής της έκθεσης. Οι τράπεζες παραμένουν μεν σημαντική πηγή χρηματοδότησης ε, εμπορικών ακινήτων στις περισσότερες χώρες της Ένωσης, ωστόσο οι μη τραπεζικοί φορείς και οι διεθνείς επενδυτές διαδραματίζουν άλλο και μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά αυτή σε σχέση με το τι γινόταν προκρίσει. Οι ασφαλιστικέ επιχειρήσεις, ε, τα συνταξιδοτικά ταμεία, τα επενδυτικά ταμεία διακρατούν πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό ομολόγων εμπορικών ακινήτων. Το μεγαλύτερο μερίδιο, όλο και μεγαλύτερο μερίδιο συνοριακής και μη τραπεζική χρηματοδότηση εμπορικών ακινήτων έχει και θετικέ πτυχέ. Συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το συνολικό επιμερισμό κινδύνου, καθότι οι απώλειες, οι ζημίες εμπορικών ακινήτων ε, επιμοιράζονται σε διάφορες φορείς και χώρες. Επίσης, σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στο εγχώρια χρηματοπιστωτικό τομέα, η πρόσβαση σε ξένες τράπεζες και άλλα ιδρύματα μπορεί να φέρει άλλες πηγές, εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Επίσης, η ικανότητα προσέλκυσης ε, κεφαλαιακών ροών θα μειώσει τη διάρκεια της ύφεση και θα τονίσει, ε, θα προωθήσει μάλλον την ανάκαμψη. Βέβαια, μπορεί αυτή η μετάβαση που σας ανέφερα να ανοίξει νέες διάβλους εμπορικών, μάλλον κραδασμών στον τομέα των εμπορικών και το που μπορούν αυτό να μεταφερθούν και στο χρηματοπιστωτικό και στην πραγματική οικονομία. Μη τραπεζικοί οργανισμοί όπως είναι τα επενδυτικά τεμεία ανοιχτού τύπου μπορούν να δεχθούν πιέσεις εξόφλησης και αυτό να δημιουργήσει σε διορθώσεις των τιμών των εμπορικών ακινήτων αν χρειαστεί να πουληθούν γρήγορα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία από τις διάφορες φορές παρεσία ξένων επενδυτών για τους οποίους δεν έχουμε και στατιστικά στοιχεία επάρκη μεταξύ άλλων επίση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο γρήγορων ε, διορθώσεων των τιμών αφού μπορεί να αποφασίσουν εύνης να ε, πάρουν τα κεφάλαιά τους αν έχουν καλύτερη απόδοση αλλού σε περίπτωση που υπάρχει κάποια βεβαιότητα στην αγορά ή ε, αν θέλουν να κάνουν ε, ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Οι ξένοι επενδυτέ επίση μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο συγχρονισμό και ευπάθεια σε παγκόσμιους φορείς κινδύνου σε τους κύκλους των εμπορικών κινητών των χρόνων. Οι μακροπολιτικές αρχές που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ευπάθειες που έχουν να κάνουν τα εμπορικά κινητά, διαθέτουν διάφορα εργαλεία. Αυτά όμως ε, είναι συγκεντρωμένα στον ε, τραπεζικό κλάδο Και λίγα μόνο τέτοια εργαλεία έχουν μέχρι στιγμής εφαρμοστεί. Με αύξηση στις σταθμίσεις κινδύνου για τις εκθέσεις των εμπορικών ακινήτων είναι το πλέον εφαρμοζόμενο μέτρο. Έχουν επίσης σε τρεις χώρες εφαρμοστεί μέτρα για τις εκθέσεις εμπορικά κίνητα ε, τα οποία βασίζονται στο δανειολήπτη. Κάποιες χώρες επίσης έχουν κάποια αποθέματα ασφαλείας ε, μακροπολιτικής εποπτείας όπως είναι απόθεμα ασφαλείας συστημικών κινδύνων ή το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας κεφαλαίου για την αντιμετώπιση των ευπαθειών που σχετίζονται με τα εμπορικά κίνητα. Ο ξανόμενο ρόλο των μη τραπεζικών ιδρυμάτων για τη χρηματοδότηση εμπορικών ακίνητων επιβεβαιώνει την ανάγκη να υπάρξουν ενδεδειγμένα εργαλεία μακροπροληπτικής εποπτείας που θα καλύπτουν όλα τα τμήματα του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου συνεχίζει να εργάζεται για την ανάπτυξη μακροπροληπτικών πολιτικών πέραν του τραπεζικού τομέα. Το SRB σήμερα λοιπόν δημοσιεύει σχετική έκθεση για το πώς μπορεί να ενισχυθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ε, ασφαλιστικές εταιρείες, για τους ασφαλιστές. Ένας υγιής ε, ασφαλιστικός κλάδος συνεισφέρει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αναλαμβάνοντας κινδύνους οι ασφαλιστές ε, έρουν το ενδεχόμενο μεγάλων ζημιών για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις και επίσης με το συνδυασμό μακροχρόνια αποταμίευση και επενδύσεων συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, η συμπεριφορά των ασφαλιστών μπορεί να οδηγήσει και στην ενίσχυση των ε, τροτών σημείων του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πιστεύει λοιπόν το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου πως θα πρέπει οι αρχές να έχουν στη διάθεσή τους ε, μια ενδεδειγμένη εργαλειοθήκη μακροπροληπτικής εποπτείας για να αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων στον τομέα των ασφαλίσεων, πέραν των μεμονωμένων ιδρυμάτων. Εν συντομία θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιε από τι βασικέ μα προτάσει. σχετικά. Πρώτον, οι αρχέ θα πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν αύξηση στο κεφάλαιο και περιορισμού στα μερίσματα σε όλο το μήκο και πλάτο τη αγορά. Έτσι θα μπορούν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των ασφαλιστών αν δεν είναι θετικέ οι εξελίξει αγορά. Αυτέ οι κεφαλαϊκέ αυξήσει θα μπορούσαν να στοχεύουν συγκεκριμένε δραστηριότητε ή φορεί. Επίση, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χρειαστεί. Μάλλον να θελήσουν κάποιοι ε, κάτοχοι ασφαλιστηρίων να τερματίσουν ε, τα ασφαλιστικά συμβόλαια σε μεγάλους αριθμούς και έτσι θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας για τους ασφαλιστές. Θα πρέπει να μπορούν να προστατέσουν τις χρηματαγορές αλλά και τους ίδιους τους ασφαλιζόμενους οι αρχές. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, τι θα μπορούσε να βοηθήσει να μην μπορούν προσωρινά, παραδείγματο χάρη, οι κάτοχοι ασφαλιστήρων να το διακόψουν, να το λήξουν. Το είχα συζητήσει και κατά το παρελθόν. Συγκεκριμένα είχα προτείνει ένα αντίστοιχο εργαλείο για τα επενδυτικά ταμεία. Μακροπροληπτική εργαλειοθήκη στους ασφαλιστέ. ίσως θα έπρεπε να περιλαμβάνει και κάποια αντικυκλικές, κάποιες αντικυκλικές κεφαλαικές απαιτήσει ε, κειμενόμενου χρόνου, ώστε να μην έχουν τόσο κίνητρο να πουλήσουν σε περίπτωση ύφεση ε, τα περιουσιακά στοιχεία και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει να μην υπάρχουν ε, ευπάθειες στον τομέα μεγαλύτερες, αυξάνοντας τις κεφαλικές απαιτήσει όταν είναι θετικές οι προοπτικές, οι οικονομικές. Επίσης, καλό θα ήταν ε, κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούνται στον τραπεζικό τομέα να επεκταθούν και στους ε, ασφαλιστές που δραστηριοποιούνται σε ανάλογες δραστηριότητες, όπως στεγαστικά δάνεια ή χρηματοδότηση εμπορικών ακινήτων. Φυσικά και εδώ χρειάζεται να γίνουν ακόμη περισσότερα. Θα πρέπει να δούμε πώ θα τα προσαρμόσουμε συγκεκριμένα αυτά τα εργαλεία, τι κατόφλια θα πρέπει να εφαρμόζονται, πώ θα πρέπει να ενταχθούν στην υφιστάμενη νομοθεσία τα εργαλεία αυτά. Το Συμβούλιο στην Κοκκινή θα συνεχίσει να τα συζητά αυτά τα θέματα και θα συνεισφέρει και στην αναθεώρηση της δεύτερης οδηγίας ε, περί χρεοκοπίας ε, ή φερεγγιότητας, το Solvency 2, βοηθώντας την Επιτροπή να αποφασίσει ποια θα είναι η μελλοντική μορφή του ρυθμιστικού πλαισίου για τους ασφαλιστές. Σας ευχαριστώ και είμαι στη θέση σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημαντική αυτή παρέμβαση. Σταθήκατε σε ένα ζήτημα το οποίο και τώρα αλλά και ε, στο επόμενο διάστημα θα απασχολήσει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας. για το θέμα της φερεγγιότητας λοιπόν. Ο κύριος Λάγκε παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω μια ερώτηση σε σχέση με τα συνταξιδοτικά ταμεία στο πλαίσιο των συνομιλιών του Εμμυρδίου ε, έχουμε τριμερή διάλογο για την συμπερίληψη των συνταξιωτικών ταμείων στο σύστημα αυτό της εποπτείας. Η Κομισιόν μείνεται εδώ και 8 χρόνια με κάθε δυνατό κόλπο ο όγκος είναι πάνω από 3, 3 εκατομμύρια ευρώ στις τρεις μεγαλύτερες χώρες. Το ερώτημά μου λοιπόν έχει δύο σκέλη. Πρώτον, η ΕΚΤ ακόμα δεν έχει εκφραστεί επισήμως πώς κρίνεται την συμπερίληψη των συνταξιδοτικών ταμείων ε, στον κανονισμό περί παραγόγων τον ΕΜΙΡ. Δεύτερον, τα συστήματα που αφορούν τις ε, τρίτες χώρες. Εάν έρθει το Brexit, ε, το οποίο μόνο αναφερθήκαμε μέχρι τώρα, το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλιστούν ακριβώς αυτά τα CCP. Κατά την άποψή μου θα πρέπει η ευθύνη να έρθει στην Ευρωζώνη, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει κάποιο μεταβατικό καθεστώς με τη Μεγάλη Βρετανία που είναι ο μεγαλύτερος τέτοιος χώρος και το άλλο θέμα αφορά τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο μέσω κύβερνο επιθέσεων λοιπά στον χώρο αυτόν. Αν δείτε παραδείγματο χάρη ε, τι έγινε με το έξω που είχαμε απώλειες φόρων δισεκατομμυρίων έχω σοβαρές επιφυλάξεις για το αν είμαστε προετοιμασμένοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα συνταξιοδοτικά ταμεία το Συμβούλιο συστημική ε, σταθερότητας έχει πει ότι δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εξαίρεση και θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Ναι, σα ευχαριστώ. Για το Brexit είναι δύσκολο ε, να πούμε εμείς δεν είμαστε στις διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι περίπλοκες και κάποιες πτυχές θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες εβδομάδες οπότε ακόμα δεν είμαστε σε θέση να πούμε το τι θα συμβεί αλλά εάν έπρεπε να μαντέψουμε το προσεχές μέλλον από τις ε, πρόσφατες εξελίξεις είναι σαφές ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει αποφασιστικότητα να αποφευθεί η υλοποίηση κινδύνων ε, χρηματοπιστωτικής ε, σταθερότητας. Δηλαδή είτε θα βοηθηθεί ο ιδιωτικός τομέας να αντισταθμίσει την κατάσταση ή όπως έκανε η Κομισιόν ότι θα υπάρξει μια πολιτική, μια δήλωση ότι δεν θέλω υπάρχουν τέτοια κίνδυνοι. Τώρα για την τελευταία σας ερώτηση. Γνωρίζετε ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένα θέμα το οποίο πλέον αποτελεί αντικείμενο προσοχή σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω οι G20 ή οι G7 μίλησαν για τον πιο σημαντικό κίνδυνο στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οπότε το σύμφωνο χρηματοπιστωτικών κινδύνων αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο για να διευκολυνθεί οι συζητήσεις ε, και ακριβώ ε, η γνώση μεταξύ των ε, μελών. Και ακριβώς ε, εστιάζουμε τώρα πιο πολύ στα ασθενέστερα σημεία. Και εστιάζουμε ακριβώς στις εποπτευόμενους φορείς που έχουν βρει τα μέλη μας και να διακρίνουμε τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί το κάθε κράτος μέλος για να βρει και να αξιολογήσει τις αδυναμίες γιατί δεν κάνουν όλοι το ίδιο έχουν ε, διαφορετική μεθοδολογία και διαφορετικέ αναφορές ε, των αδυναμιών οπότε προσπαθούμε τώρα να σχηματίσουμε μια άποψη για τις ε, στάθειες εκείνες, τις αδυναμίες εκείνες που αφορούν ολόκληρο το σύστημα και τους διάβλους διάδοσης που είναι ηλεκτρονική και οπωσδήποτε αυτό θα βρεθεί στις ε, συζητήσεις μας σε τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτιμούμε το ότι η ΕΚΤ έχει την ίδια θέση με μας σε αυτές τις συζητήσεις και βεβαίως ε, Εκτιμήσαμε ακριβώ ε, την ε, ανακοίνωση στα μέτρα αυτά που μας υπενθύμησαν ότι οι ισοδύναμες αποφάσεις μπορούν να ληφθούν πάρα πολύ γρήγορα αν υπάρξει ανάγκη λαμβάνοντας υπόψη βεβαίω ότι θα προτιμούσαμε να μην χρειάζεται να δούμε αν επαρκούν τέτοια μέτρα Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με την ψηφοφορία στην Βουλή των Κοινοτήτων. Υπέρ Βανσμπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στα εμπορικά ομόλογα. Ήταν ένα από τα θέματα που είχαμε εξετάσει με το ESRB όταν ε, είχαμε συνδράμει και εμείς το έργο σας. Κατανοούμε ότι ανάλογα και με τα επιτόκια μπορεί να υπάρχει ε, ένα μικρό μερίδιο της αγοράς που θα μπορούσε κανείς να εκμεταλλευτεί. Υπάρχουν ε, φορείς Τη αγορά χρηματοοικονομικών που παρεμβαίνουν σε αυτά τα εμπορικά ομόλογα. Θεωρείτε όμως ότι πρέπει ε, να ε, εξελίξουμε περαιτέρω την νομοθεσία ή απαιτείται απλώς εποπτεία και παρακολούθηση σε διαφορετικό όμως επίπεδο. Τι επιθυμείτε να κάνετε. Αν ε, επιθυμείτε αλλαγή της νομοθεσία, θεωρώ ότι υπάρχει μια δυσκολία γιατί αφενός έχουμε ε, την νομοθεσία για τον τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης ε, των ομολόγων αυτών από τον τραπεζικό κλάδο, αλλά υπάρχει και η νομοθεσία για τα εμπορικά ομόλογα αυτά καθ' αυτά. Έχετε λοιπόν προσδιορίσει χώρες όπου η νομοθεσία ε, ευνοεί τη δημιουργία αυτού του μεριδίου της αγοράς ή όχι. Μετά, είπατε ότι πρέπει να έχουμε πιο μακροπροληπτική προσέγγιση ε, για τους ασφαλιστές. Πού θεωρείτε, σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να επιληθεί ε, το ζήτημα, να περιμένουμε συστάσεις του ESRB ή νομίζω ότι κάπου αλλού θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα. Ε, ευχαριστώ. Για το δεύτερο στοιχείο που αναφέρατε για τους κινδύνου που έχουν να κάνουν όμως και πάλι με τον ε, τομέα των εμπορικών ακινήτων. Είπα και πριν ότι επειδή είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος και μεγάλη η ε, διασύνδεση, απαιτείται μεγάλη προσοχή. Βασικός, ε, βασική αιτία των ευπαθειών που έχουμε εντοπίσει εμείς τουλάχιστον σε αρκετές χώρες είναι η προσπάθεια αναζήτησης απόδοσης από τους επενδυτές. και αυτό οδηγεί σε εξαιρετικά υψηλές ε, εκτιμήσεις ε, για τα εμπορικά ακίνητα, ιδίως στην πρωτογενή αγορά. Και έτσι ε, γίνονται έτσι πιο... Αυξήνεται ο κίνδυνος ανατιμολόγησης και έτσι αυξάνεται και ο κίνδυνος πιθανών κραδασμών και ευπαθειών. οι τράπεζες ε, πράγματι δεν ε, εκτίθενται σε αυτό το κίνδυνο. Είναι ο μη τραπεζικό κλάδος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πώς συνδέονται λοιπόν αυτές οι μη τράπεζε με το τραπεζικό σύστημα και μέσω αυτού με την πραγματική οικονομία. Γι' αυτό και το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και εν γέννη όλες ε, οι αρχές μακροπροληπτικής πολιτικής και σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΚΤ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύτερο μέσο ε, εργαλείων, μια μεγαλύτερη εργαλειοθήκη που να μπορεί να επεκταθεί πέραν του τραπεζικού κλάδου και στο μη τραπεζικό. Θα έπρεπε επίσης να υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης ορατότητας αυτών των ε, επενδυτών για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την διασύνδεση αυτών των ε, μη τραπεζών με το υπόλοιπο σύστημα. Όπως λοιπόν και γενικότερα στο ε, σύστημα θα πρέπει να καταβάλουμε κάποιες προσπάθειες για να προστατευτούμε από τέτοιους κινδύνους. Με ρωτήσατε για ε, την μίσθωση χρόνου με το ακινήτων ε, και δεν το γνωρίζω τώρα συγκεκριμένα. Πρέπει να το διερευνήσω περαιτέρω. Αν ε, βρω κάποια διαφορετική απάντηση θα σας την διαβιβάσω γραπτός. Πρέπει λοιπόν να διευρύνουμε την μακροπροληπτική εργαλειοθήκη για να συμπεριληφθεί εδώ και ο μη τραπεζικό κλάδο αλλά και ο ασφαλιστικό κλάδο. Συμφωνώ απολύτω. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά. Όμως εδώ το, το έργο μας είναι πιο απλό καταρχήν, γιατί το εύρος των φορέων και των οντοτήτων είναι μικρότερο. Ενώ στον μη τραπεζικό κλάδο τα πράγματα είναι πιο δύσκολο να τα ορίσει κανείς. Ναι, αλλά θεωρείτε ότι το ESRB είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να αναλάβει τον μακροπροληπτικό κίνδυνο του ασφαλιστικού κλάδου, γιατί μετά θα πούν ότι δεν εκπροσωπούνται επαρκώς ε, στο ESRB. Όχι, εκπροσωπούνται, ε, στο ESRB, αλλά ε, το ESRB δεν είναι όργανο λήψης αποφάσεων. Έχει έναν ειδικό σχεδιασμό λοιπόν το ESRB που εστιάζει περισσότερο στην ανάλυση, ε, στις ανακοινώσεις και τις συστάσεις, όχι στην επιβολή νομοθεσίας. Οι συστάσεις μάλιστα φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματικό μέσο. Για να πετύχουμε αλλαγή πολιτική σε κάποια κράτη-μέλη από ό,τι θεωρούσαμε στην αρχή. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το ESRB θα πρέπει να έχει ε, ιδιότητε και αρμοδιότητες μακροπροληπτικής εποπτεία. Οι εθνικές αρχές και οι κεντρικέ τράπεζε είναι αυτές που έχουν αυτή την αρμοδιότητα. Και το θεσμικό όργανο το οποίο όλοι θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί αυτομάτως είναι ο ΑΙΟΠΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλής και Πολιτικών Συντάξεων. Ο κύριος Τραμόσα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Ντράγκη, έχω δύο ερωτήματα. Μιλήσατε για τον τομέα των ακινήτων. Για τα κόκκινα δάνεια, καθώς πολλά προκύπτουν από φούσκες, μετά από τον τελευταίο επεκτατικό επιχειρηματικό κύκλο πριν από 10 χρόνια. Εξετάζουμε τώρα μια πρόταση κανονισμού για τα ε, μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το Συμβούλιο έχει, συνηθίσει, έχει συμφωνήσει ήδη επί γενικής θέσης και φαίνεται ότι θα περάσει ο φάκελος. Η προσέγγιση του Συμβουλίου προβλέπει ένα ομοιόμορφο χρονοδιάγραμμα που θα εφαρμόζουν οι χρηματοοικονομικοί φορείς ε, για την δημιουργία των ε, ασφαλιστικών δικλείδων. Εσείς δεν φοβάστε κάποιο ασύμετρο κρατασμό στα κράτη-μέλη γιατί κάποιες ε, τράπεζε μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην δημιουργία αυτών των δικλείδων. Και μετά, Τις περασμένη εβδομάδα έχουμε κάνει μια ε, δύσκολη συζήτηση σε αυτή την Επιτροπή για την, ε, την έννοια της, ε, του failing ή του likely to fail. Ο επικεφαλής του ESRB είπε πριν από ένα μήνα ότι αυτός ο ορισμός είναι εξαιρετικά δύσκολος η κυρία Νουή όμως τη ρώτησα την περασμένη εβδομάδα και μας είπε ότι θεωρεί ότι είναι αρκετά σαφή ο ορισμό. Εσείς θεωρείτε ότι είναι αρκετά σαφής ο ορισμός για τις προβληματικές τράπεζες ή αυτές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Το δεύτερο ερώτημα είναι πιο εύκολο να απαντήσουμε. Ό,τι σας έχει πει η κυρία Νουή ισχύει και είναι ορθό. Εκείνη είναι αρμόδια. Αν ο SSM έχει συμφωνήσει με αυτόν τον ορισμό, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για το άλλο ερώτημα, τι εννοείται με backstops, την απόρριψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή την κάλυψή τους μάλλον. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω με ένα θετικό μήνυμα, ότι έχει σημειωθεί πρόοδος ότι φορά την μείωση των κόκκινων δανείων. Ήταν 7,5% στις αρχές του 2015 και έχουμε πέσει στο 3,6% στο δεύτερο τρίμηνο του 2018. Έχουν πέσει λοιπόν σημαντικά στα αθρηστικά στοιχεία. Βέβαια το πρόβλημα είναι με τα κόκκινα δάνεια ότι τα αθρηστικά στοιχεία λένε λίγα. Όμως γενικά έχουμε μια καθοδική τάση σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, ο συντελεστής κάλυψης είναι 46% το δεύτερο τρίμηνο του 2018 και ήταν 46,5% στο πρώτο τρίμηνο. Υπάρχει βελτίωση, λοιπόν, αλλά δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα. Και πάλι ε, υπάρχει αυτό το ζήτημα του στελιστή κάλυψης. Το ESRB εργάζεται άοκνα σε αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα και υπάρχει ένα εξαιρετικό έγγραφο που δημοσίευσε η Συμβουλευτική ε, Επιστημονική Επιτροπή για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ε, για τα ενολογικά θεμέλια μιας μακροπροληπτικής προσέγγισης σε αυτό το ζήτημα. Συνεχίζουμε να το επεξεργαζόμαστε λοιπόν αυτό και καταβάλουμε προσπάθειες για να εντοπίσουμε τις ευπάθειες που προκύπτουν από αυτά. Είναι ένα βαρύδι για το τραπεζικό σύστημα, είναι σαφές. Εάν δεν είχαμε κόκκινα δάνεια ή αν ήταν χαμηλότερος συντελεστής, θα μπορούσε και το τραπεζικό σύστημα να δίνει μεγαλύτερες πιστώσεις και να τοποκρίνεται περισσότερο στην ευρύτερη οικονομία. Αυτό είναι σαφές. Τώρα, κάποιε χώρε προσπαθούν να συνδέσουν την πρόοδο στο μέτωπο αυτό των κόκκινων δανείων σε σχέση με την πρόοδο που σημειώνεται στην ε, Τραπεζική Ένωση ότι όλα αυτά συνδέονται με τα κόκκινα δάνεια. με προτάσεις ε, που δείχνουν ότι πρέπει να επιτευθούν ε, ποσοτικοί στόχοι για τα κόκκινα δάνεια εάν θέλουμε να συμφωνήσουμε επί περαιτέρω βημάτων στην Τραπεζική Ένωση. Αξίζει ε, και χρήζει στήριξη σε αυτή η προσέγγιση. Δεν είμαι σίγουρος ότι ε, αυτή η αναγνώριση στόχων ε, παντού είναι η καλύτερη προσέγγιση. Αυτό που έχει κάνει ο SSM είναι ότι έχει ε, συγκεκριμένες προβλέψεις και προσδοκίες και έχει έναν πολύ αποτελεσματικό διάλογο με πολλές μεμονωμένες τράπεζες και οι δύο πλευρές προσπαθούν να θέσουν στόχους μία τράπεζα τη φορά. Και αυτή η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα επιτυχής. Τώρα, κατά πόσο οι τιμές που αναφέρονται εκεί δεν είναι ρεαλιστικές, δεν το νομίζω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, εργαζόμαστε πάνω στο θέμα αυτό του χρονοδιαγράμματος και θα δούμε προσεχώς τις ε, τροπολογίες. Βεβαίως το ερώτημα του κυρίου Μόζε αφορούσε ε, τον κίνδυνο μιας αυτόματης τέτοια παροχής ε, στον πυλώνα ένα που ίσως κινδύνευε να ενισχύσει τις τάσεις της οικονομικής συγκυρίας. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι το Συμβούλιο και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε στο Κοινοβούλιο θα αυξήσει ακριβώ ε, την πρόβληψη αλλά όχι υπερβολικά γιατί αυτό κατά την άποψή μου θα μπορούσε πράγματι να δημιουργήσει προβλήματα με το να ενισχύσει τις ε, κύκλικες ε, τάσεις είναι λοιπόν αποτελεσματικό ενισχύει τον πυλώνα 1 ενώ ο πυλώνας 2 που αφορά την κάθε τράπεζα ξεχωριστά εξαρτάται και από την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματο και το πλαίσιο. Κύριος ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Θεωρώ λυπηρό και αδιανόητο το ότι έχουν έρθει τόσοι ε, λίγοι συνάδελφοι στον ε, νομισματικό διάλογο με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το λέω ανοιχτό, ανοιχτά είναι αδιανόητο εγώ ήμουν πάντα εδώ από την εποχη Ντουζενμπερκ. Ντούζεμπεργκ. Έχω λείψει δύο-τρει φορές, αλλά σε 80 νομισματικούς διαλόγου δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Προφανώ εξαιρούνται οι παρόντε. Ε, πραγματικά δεν ξέρω. Φαντάζομαι καταρτίζονται οι λίστες οι προεκλογικές, αλλά δεν είναι δυνατόν να μιλά εδώ πέρα μόνος του πρόεδρο τη. της ΕΚΤ. Δεν έθεσα όμως το αγαπημένο μου ερώτημα, κύριε πρόεδρε το θέμα ακριβώς της αξιολόγησης κινδύνου των ε, κρατικών ομολόγων. Γνωρίζω τους ε, κινδύνους ε, εάν υπάρχει κάποια αξιολόγηση κινδύνου. Γνωρίζω ότι αξιολογούνται τα τραπεζικά ιδρύματα, βλέπουμε την άνοδο των επιτοκίων και υπάρχει οπωσδήποτε και η αναλογική κερδοσκοπία. Από την άλλη πλευρά όμως εδώ και 10 χρόνια έχουμε την συζήτηση στην Επιτροπή της Βασιλείας για τον διαχωρισμό τραπεζών και κρατών και αυτό στην Νότια Ευρώπη τελικά οδήγησε στο ότι αυξήθηκε το μερίδιο των κρατών στις τράπεζες. Ε, υπάρχουν πλέον εκτίματα και μειονεκτήματα. Βλέπετε κάποια διέξοδο από αυτό κύριε Πρόεδρε όσον αφορά την ε, αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων. What is the last question you asked? Α, τελευταία ερώτηση που κάνατε. Υπάρχει μια, κάποια πρόταση για να βγούμε από αυτήν την ε, κατάσταση της μη αξιολόγησης του κινδύνου αλλά και των προβλημάτων που θα παρουσίαζε το να το κάνουμε τώρα. Υπάρχει κάποιο άλλο μέσο μακροπρόθεσμα, τι μορφή θα μπορούσε να έχει μια λύση. Σας ευχαριστώ. Ε, πράγματι υπήρχε, έχετε δίκιο, μια συζήτηση που τράβηξε πάρα πολύ στην Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία τελικά αποφάσισε να μην κάνει τίποτα, γιατί το δημόσιο χρεο αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Στον υπόλοιπο κόσμο θεωρείται ότι δεν έχει κίνδυνο το δημόσιο χρεο οπότε δεν ε, ζητάνε από τι τράπεζε να αξιολογήσουν ε, το σχετικό ρίσκο. Βεβαίω ο λόγο είναι ότι πάντα υπάρχει η κεντρική τράπεζα για να τυπώσει χρήματα, για να στηρίξει το δημόσιο χρέο Εάν χρειαστεί αυτό, εξυπονοείται. Τώρα, εάν ισχύει, αν συμβαίνει ή όχι, είναι κάτι το διαφορετικό. Ε, στην περίπτωσή μας, ε, στην περίπτωση της Ευρωζώνης, ανακαλύψαμε ότι το δημοσιοχρέος ε, δεν είναι απαλλαγμένο κίνδυνο. οπότε στο βαθμό αυτό το να πούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε ως κάτι το οποίο παρουσιάζει κίνδυνο στον ισολογισμό των τραπεζών ισχύει. Το, το πώς θα γίνει αυτό. Η απάντηση δεν είναι απλή γιατί ακριβώς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μέτρα τιμών και όχι ποσοτικές οροφές. Ταυτόχρονα, και αυτό ήταν το ζήτημα στην Επιτροπή της Βασιλείας, υπάρχει το θέμα των ίσων όρων ανταγωνισμού. Εάν ζητήσουμε από τις τράπεζες της Ευρωζώνης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν τέτοιες αξιολογήσεις ε, κινδύνου σημαίνει ότι οι επενδύσεις σε κάποια στοιχεία είναι πιο ακριβές από ότι για τις ε, τράπεζες που είναι σε άλλα μέρη του κόσμου. Οπότε υπάρχει το θέμα των ίσων όρων του ανταγωνισμού. Γενικότερα θεωρώ ότι οι δράσεις ε, προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν κατά νου τις ε, πιθανές επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε διάφορα μέρη της Ευρωζώνης σε διάφορα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να είναι και μέρος ενός ευρύτερου πακέτου, όπου εάν κάποιος χάσει την ευελιξία που μπορεί να παρέχει το τραπεζικό σύστημα στην στήριξη του χρέους και των ελλημάτων, θα ήθελε να δει πρόοδο σε άλλα τμήματα του συνολικού πακέτου της ενίσχυσης ε, της ΟΝΕ. Οπότε αντικειμενικά είναι δύσκολο να γίνει η συζήτηση και υπάρχει και κάτι άλλο, μια άλλη πτυχή. Όταν μια χώρα όπως λένε χρεοκοπήσει δεν έχει διαφορά αν μία τράπεζα έχει πολύ λίγο δημόσιες, ε, δημόσιο χρέος όλες οι τράπεζες ε, θα υποφέρουν είτε έχουν ε, πολλά ή λίγα κρατικά ομόλογα. Οπότε πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση γιατί δεν είναι απαλλαγμένα κινδύνου τα κρατικά ομόλογα και ταυτόχρονα είναι και περιπλοκή. Αλλά δεν θα πρέπει να αγνοούμε την πραγματικότητα. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι, πολύ πλόκο. Είναι το θέμα. Ιδίω αν ληφθεί υπόψη ότι ζητείται και ο από τον ίδιο κανονισμό να έχουν ε, οι τράπεζες ε, αυτά τα high liquid ε, risk assets στον προπολογισμό τους. Και αν δεν το έχουν, it's Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. και φαύλος κύκλος. Ίσως θα έπρεπε να μπει σε ένα ευρύτερο πακέτο. Έχετε δίκιο. Περιβάνς Μπερές. Ευχαριστώ. Για πέμπτη, αλλά τελευταία φορά σήμερα θα πάρω το λόγο αυτή τη φορά σε σχέση με το Συμβούλιο Συστημικού Κατά κάποιο τρόπο αυτή την ε, μακροπροληπτική εποπτεία, την τραπεζική, εσείς ε, την ε, θεσμοθετήσατε. Σήμερα έχουμε το θέμα πώς θα διαρθωθεί μαζί με την άλλη σας ιδιότητα. Ως συνεισηγητής της αναθεώρησης της διακυβέρνησης του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, θέλω να μου πείτε πώς αξιολογείτε εσείς το σημερινό σύστημα διακυβέρνησης. Από τη μια πώς χρησιμοποιείται και αξιοποιείται την Επιστημονική Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα και το Συμβούλιο πώς συνεργάζονται. Όταν δημιουργήσαμε αυτή τη μακροοικονομική εποπτεία μέσα στην κρίση γίνανε κάποιες ε, πολύ οδυνηρές συνειδητοποιήσεις τότε για το τραπεζικό τομέα, σήμερα τα λέτε τα ίδια για τον ασφαλιστικό κλάδο. Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση και τον αντίκτυπο για τη δημοσιονομική πολιτική. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η συνολικότερη άποψη για τους μακροοικονομικούς κινδύνους. Yes, I, I, I completely, completely agree. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας. Βήμα που το πάμε εδώ. Καταρχάς, να δούμε πόση δουλειά έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από το Συμβούλιο και τι μεγάλο πεδίο εφαρμογή έχουμε καλύψει και φαίνεται και από τη σημερινή συζήτηση. Έχει δουλέψει καλά το Συμβούλιο. Βέβαια, εγώ ε, δεν είμαι και ο πιο αντικειμενικό ε, παρατηρητής. Αλλά νομίζω και εσείς θα δεχτείτε ότι πολύ αποτελεσματικά αντόπισε κινδύνους, ευπάθειες, ε, έκανε συστάσεις, προειδοποίησε, έκανε υποδείξεις κτλ. Σε συμμόρφωση προς την εντολή που του είχε δοθεί πριν από αρκετά χρόνια. Τώρα, μετά, πριν δύο χρόνια νομίζω, τρία, ετέθη το θέμα ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εποπτικού, ε, Συστημικού Κινδύνου να είναι στην διάδρα με, τον Ευρωπαϊκό, με την Ευρωπαϊκή Κεντρικά Τράπεζα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια σύγκρουση. Και όσοι ρώτησα, ούτε αυτοί ε, μπορούσαν να εντοπίσουν σύγκρουση συμφερόντων πουθενά. Και για τον εξή πολύ απλό λόγο συμπληρώνει την πνευματική πολιτική η μακροοικονομική πολιτική. Δεν είναι κατά αυτής. Και πιο συγκεκριμένο. Πολλές φορές υπάρχει το επιχείρημα ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα οφείλεται στα χαμηλά επιτόκια που παρατείνουν τις περιόδους ρευστότητας που θα μπορούσε αυτό να σημάνει την απαρχή μιας επόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πώς απαντάμε σε αυτό εμείς από το ECBR? Η αλλαγή στην νομισματική πολιτική, ακριβώς λόγω αυτού, δεν νομίζουμε ότι θα έχει νόημα. Γιατί θα έθετε σε κίνδυνο την ανάκαμψη. Πολύ απλά. Αν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση εδώ είναι πρέπει να θεωρηθούν οι κατάλληλες ε, μακροπροληπτικές πολιτικές. Και πώς λοιπόν τελικά αλληλοσυμπληρώνονται οι νομισματικοί με την μακροοικονομική πολιτική, άρα δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ίσα ίσα. Δημιουργούνται συνέργειες και το υπονοήσατε νομίζω στην ερώτησή σας. Άρα, συμπερασματικά δεν είναι δική μου δουλειά να συζητήσω τη κυβέρνηση, γιατί είμαι αντικείμενο αυτή τη συζήτησης, αλλά νομίζω ότι η διακυβέρνηση του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου έχει λειτουργήσει καλά και όσοι εργαζόμαστε στο πλαίσιο αυτού του Συμβουλίου δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι στη διακυβέρνηση. Φυσικά μπορεί να βελτιωθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία, η υποβολή αναφόρων φυσικά και είμαστε διατεθειμένοι να φέρουμε σε πέρασα όλες τις απαιτούμενες βελτιώσεις. αλλά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να μπούμε σε ένα μονοπάτι που θα δημιουργούσε πλουραλισμό, πολυφωνία στις έξωτερα αναφορές από πλευρά Συμβουλίου ή εδώ παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι φυσιολογικό να οδηγήσει σε διαστάσεις απόψεων και να πλήξει τη φήμη και των δύο θεσμών αυτό. Να προσθέσω ότι λέει η κυρία Μπέρες, ότι ο Βέρνερ Λάγκε που είπε ότι είναι ένα σκάνδαλο που δεν είμαστε σήμερα περισσότεροι εδώ, με βρίσκει απολύτω σύμφωνο. Όταν καθορίστηκε αυτό ο, παγιώθηκε αυτός ο διάλογος, ο νομισματικός, ήμασταν ε, και οι δυο μας εδώ και πραγματικά σίγουρα μπορεί κάποιοι να ασχολούνται με τα ψηφοδέλτια, αλλά δεν, δεν είναι δυνατόν να είμαστε τόσοι λίγοι εδώ. Ο Πρόεδρος, συμφωνώ απόλυτα. Ένα τελευταίο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της συνταλλαγής απόψεων έχουμε συζητήσει πολλά θέματα ασφάλισης, δημοσίου χρέους, μη εξυπηρετουμένων δανείων. Να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Δεδομένου ότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είδαμε και δικαστικές αποφάσεις ότι ο δανεισμός μόχλευσης και άλλα προϊόντα που ξέρουμε ότι εν μέρη ευθύνονται για την ε, οικονομική κρίση, χρησιμοποιούνται και πάλι. Ποια είναι η δική μας εκτίμηση. Βρισκόμαστε εμείς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουμε τους δικούς μας κανόνες, είμαστε πλέον ασφαλείς. μπαίνουν αυτά τα στοιχεία στους ολογισμούς των τραπεζών, υπάρχει πρόβλημα με το μη τραπεζικό κλάδο που συνδέεται τελικά και με τον τραπεζικό. Τα όσα κάνουμε και εμείς και εσείς φτάνουν. Υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι που θα πρέπει να παρακολουθούμε πιο στενά 10 χρόνια μετά την υπόθεση με τη Lehman Brothers. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όντω ε, μια κίνηση προ την αντίθετη κατεύθυνση σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Δηλαδή, προχωρούμε σε απορρίθμιση. Είτε αυτό προέκυψε μέσω της νομοθετικής διαδικασίας ή μέσω της αλλαγής από τους υποπτικούς μηχανισμούς, είτε όπως είπατε και από δικαστικές αποφάσεις. Μία συγκεκριμένα αφορούσε την ε, συγκράτηση ε, κινδύνου, η διατήρηση κινδύνου σε συγκεκριμένα ε, προϊόντα. Είδαμε λοιπόν ότι κάποια, τα οποία δεν τα είχαμε ξανακούσει μετά την οικονομική κρίση, CDOs, CLS, τώρα τα αρχίζουμε να τα ακούμε πιο συχνά πάλι. την Ευρώπη τώρα. Το πρόβλημα για κίνδυνος ποιο είναι, ότι ψάχνουμε να βρούμε αποδόσεις και μπορεί να επαναληφθούν ε, οι αρνητικές αυτές συμπεριφορές που ε, τελικά μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Δηλαδή πολλές, ε, πολλοί φορείς και τράπεζες και μη τράπεζες ψάχνουν υψηλέ αποδόσεις και έτσι πέφτουν σε αυτά που αποκαλούμε τοξικά προϊόντα που τελικά ήταν ε, ο βασικός μοχλός ε, της κρίσης ε, στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση και χρονική συγκυρία, η έκθεση σε αυτά τα νέα προϊόντα σε μεγάλο βαθμό αφορά τις μη τράπεζες. Έτσι έχουμε και πάλι λόγο να έχουμε μεγαλύτερη ε, κάλυψη και του μη τραπεζικού κλάδου, δηλαδή να επεκταθεί η εργαλειοθήκη μας για να καλύψει και τον μη τραπεζικό κλάδο, αλλά και να παρακολουθούμε την έκθεση των τραπεζών μας σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Να δούμε αν αυτή τη στιγμή ή στο μέλλον αυξηθεί η έκθεσή μας, ε, κάτι το οποίο θα μας ε, ανησυχήσει στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και είναι κρίμα πραγματικά ότι δεν ήρθαν περισσότεροι βουλευτές παρά το ότι όλοι αιρετοί είμαστε και αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται κανείς τη χώρα του σε κρίσιμε στιγμέ. Ε, νομίζω ότι πολλά από τα ζητήματα που συζητάμε είναι πολύ σημαντικά και ελπίζω να έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και να αποφύγουμε κάποιους ε, κινδύνους μετά από τόσες προσπάθειες που κάναμε να αφήσουμε σκληρονομιά ένα ε, ανθεκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο χωρίς ε, παραθυράκια τα οποία θα υπονομεύσουν όλη αυτή τη δουλειά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τα πολύ σημαντικά πράγματα που είπατε για τον πολύ ενδιαφέροντα διάλογο. Λοιπόν, τελειώσαμε το θέμα αυτό. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε στις 6 η ώρα.